Uh, Καλημέρα σε όλους σας. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Θα ήθελα να, καλωσορίσω, να σας καλωσορίσω στην ε, δεύτερη μέρα των, ε, της συνάντησής μας. Πολύ σημαντική συνεδρίαση πιστεύω. Λοιπόν, σας παρακαλώ να καθίσετε Λίγη ησυχία παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην, ε, στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης, της, μάλλον στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας. Έχουμε πολύ δύο σημαντικά θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Καταρχάς, η σύναψη δημόσιων συμβάσεων είναι μια μισή ώρα που θα αφιερώσουμε σε αυτό το θέμα. Βλέπετε πόσο σημαντικό το κρίνουμε και μετά στις 10.30 θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους και πυρογνώμες Επιτροπής για ένα άλλο σημαντικό θέμα που είναι η απόσπαση εργαζομένων και σήμερα το απόγευμα η κυρία Βερνιό θα μας, δώσει, θα μας παρουσιάσει τις απόψεις της ε, για την ε, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σε με διοικητική συνεργασία. Λοιπόν, ε, καταρχάς ε, να σας πω ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για τις δημόσιες συμβάσεις. Λοιπόν, καλωσορίζω τον κύριο Ταραντέλα που είναι ο εισηγητής μας και τους κοιόδης εισηγητές από τις διάφορες ομάδες. Κάποιοι έχουν έρθει, κάποιοι όλοι, κάποιοι όχι. Λοιπόν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ε, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μάρκα Ταραμπέλα να ξεκινήσει τη συζήτηση για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η σημερινή συνάντηση και συζήτηση θα ε, εστιαστεί στα πέντε πρώτα κλάστορ των τροπολογιών, στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις, περιορισμός των εγγράφων που απαιτούνται, δηλαδή μείωση της γραφειοκρατίας, ε, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις, ε, στην αγορά των δημόσιων συμβάσεων. Ούτως ή άλλως εδώ μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα για την ε, ολοκλήρωση της ε, εσωτερικής αγοράς. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι το 19% του ΑΕΠ, όπως λέει ο κ. Μπαχνιέ. Επομένως, επηρεάζει ο τομέας αυτός τις ε, κρατικές δαπάνες, άρα πρέπει να αναθεωρηθεί ο τομέας αυτός και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, βέβαια δεν μας αφορά ακόμα, αλλά θα πρέπει να, για να επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη χρειάζονται περισσότεροι κανόνες ε, μεν, αλλά μεγαλύτερος εξυγχρονισμός, λιγότερη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να προασπίσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, θα πρέπει να σεβαστούμε κάποια κοινωνικά και περιβαλλοντικά ε, κριτήρια. Θέλω να συζητήσουμε μαζί σας, συνάδελφοι, τις τροπολογίες που υποβάλλετε, διότι κάποιες από αυτές ε, τις τροπολογίες δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες ε, ή τόσο φιλόδοξες σας θέλαμε. Ενώ άλλες αναφέρονται στις ε, τροπολογίες ε, ε, αναφέρονται συγγνώμη, στην, στους φιλόδοξους στόχους για την προστασία των κοινωνικών διατάξεων, του περιβάλλοντος κτλ. Κάτι το οποίο θέλουμε. Η εναρμόνιση των αγορών και κυρίως οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να εμφανίζονται με έναν αδιάφανο τρόπο. Το, συμφωνώ με το άρθρο 24 της οδηγίας η απλούστευση είναι ένας βασικός στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχουμε μέσω αυτής της οδηγίας. Όλοι μιλάμε για αυτήν και πρέπει να την α, ε, πετύχουμε. Αυτή η απλούστευση βέβαια δεν ελήφθη υπόψη επαρκώς και βλέπουμε ποιες είναι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί όσον αφορά τις διαδικασίες. Ε, θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα σύναψη συμβάσεων πιο απλό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, συντομεύονται και οι διαδικασίες, ε, κυρίως αν δεν έχουμε φροντίσει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ε, προϋποθέσεις. Το βλέπουμε και για, το, για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Οι αναθέτουσες αρχές βέβαια θα πρέπει να επιβάλλουν ούτως ή άλλως σε πρώτες την, τις απουστευμένες διατάξεις, άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτική και στην εφαρμοστικότητα των διατάξεων που θα υιοθετήσουμε. Τώρα, ε, οι διαδικασίες ε, μέσω διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι και αυτές ε, διάφανες. Υπάρχουν συνάδελφοι που υπέβαλαν τροπολογίες για το 24-3, δηλαδή να είναι απλουστευμένες οι διαδικασίες αλλά ευέλικτες. Κάτι άλλο είναι η, η επιλογή που πρέπει να γίνει ε, ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως ε, ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν ήταν όπως τα θέλαμε. Ε, πέντε χρόνια μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται για να συναυθεί μια δημόσια σύμβαση, Άρα αυτές οι αβέβαιες διαδικασίες μας οδήγησαν την Κομισιό να υποβάλει μια νέα πρόταση, τη συνεργασία για την ανακαίνιση, ας πούμε, ανανέωση. Υπάρχουν ε, ωραίες λέξεις βέβαια είναι αυτές, ε, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε βέβαια τον ανταγωνισμό και όταν μιλάμε για καινοτομίες και για ανανεώσεις τέλος πάντων, θα πρέπει να ε, ε, υπάρχει και μια πραγματικότητα. Ωραίες οι λέξεις, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία η οποία βέβαια άλλες φορές θα αφορά περισσότερο την καινοτομία ή ε, τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε, στις επιχειρήσεις. Αλλά κατά την άποψή μου πιστεύω ότι ο κύριος Άγγελο και ο κύριος Αρμπούρ που ε, ναι μεν <clears throat> ε, προτείνουν αυτή την συνεργασία για την καινοτομία, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε όλα αυτά να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις, να υπάρχει δηλαδή μια ενιαία γραμμή. Λοιπόν, ένα από τα σημεία κλειδιά της, ερώτησή αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές στο άρθρο 40 και στην ε, διαδικασία ε, παραγωγή, της, ε, παρα, μιας παραγωγής κοινωνικής βιωσιμότητας. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται σεβαστές και κάποιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και να μιλάμε μόνο απλώς για προϊόντα ενδυναμώνουμε την ε, στρατηγική των ε, δημόσιων συμβάσεων και αυξάνουμε την διαφάνεια στη σύναψη. Ε, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι στρατηγικής σημασίας, διότι είδα ότι μέσω κάποιων τροπολογιών εκφράζεται με κάποια καχυποψία. Η συμπερίληψη και κάποιων κριτηρίων που αφορούν κοινωνική ολοκλήρωση τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Εάν η αναθέτουσα αρχή ε, θέλει να είναι πιο φιλόδοξη, μπορούμε να τη το επιτρέψουμε. Πολλοί συνάδελφοι υποστηρίζουν και υποστήριξαν ε, την, ε, το κριτήριο της, της προσφοράς της πλέον ικανοποιητικής από την και από πλευράς ε, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, υπάρχει επίσης και μια πειθαρχία, την οποία προτείνω πειθαρχία για τις ε, υπεργολαβίες. Έχω προτείνει κάτι τέτοιο, σταδιακά βέβαια, αλλά παρόλα αυτά είναι ε, θεμελιώδης Γιατί πολλές φορές ε, τα προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις προέρχονται από μη ελεγχόμενες ε, υπεργολαβίες. Πολλοί θεωρούν ότι την υπεργολαβία δεν πρέπει να την αγγίξουμε, είναι θέμα ταμπού. Όμως εγώ θεωρώ ότι όταν χάνονται τα χρήματα είναι μέσα από μια αλυσίδα η οποία δεν ελέγχεται ε, για μια δουλειά την οποία δεν την κάνουν καλά κάποια άτομα, από κάποια άτομα τα οποία ή δεν έχουν τα προσόντα είτε έχουν ε, λάθος σύμβαση. Άρα θα πρέπει να αναφερθούμε και στην συνυπευθυνότητα αυτών που αναθέτουν ε, σε άσχετους υπεργολάβους. Η Κομισιόν στο άρθρο 62 αναφέρεται σε άλλες, άλλους φορείς λέει ότι οι αναθέτουσες αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να απαιτήσουν ε, όλοι οι οι φορείς που αναλαμβάνουν το έργο να είναι συνυπεύθυνοι. Επομένως, πιστεύω, επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα της υπεργολαβίας. Ε, και μέσω των συμβάσεων, αν θέλετε, που συνάπτει ο οικονομικός κόσμος. Τώρα, περνάω στο κλάστερ 3 ε, και 4, φτάσαμε στο επιδόρπιο, διότι ο περιορισμός των ε, εντύπων, των απαραίτητων εντύπων και το ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Ε, βέβαια, εδώ αντιμετωπίζονται τα θέματα με ένα κατακριματισμένο τρόπο, διότι οι ρήτρε εξαίρεσης δεν μπορεί να αποτρέψουν από τις δημόσιες αρχές να απαιτήσουν συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες. Λοιπόν, δεν μπορούμε το, γιατί τις ηλεκτρονικές ε, συμβάσεις να περιοριστούμε μόνο σε ένα κομμάτι της αγοράς. Επομένως, δεν πρέπει να θέτουμε περισσότερα εμπόδια από ότι να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Δηλαδή μπορεί να αναβάλουμε την εφαρμογή του για το 2017, αλλά θα πρέπει να είναι γενική η εφαρμογή. Χρειάζεται διοικητική απλούστευση και για τις επιχειρήσεις και για τις αναθέτουσες αρχές, αλλά το επαναλαμβάνουμε σημαντικά ότι αυτοί, αυτές οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις θα στεφθούν με επιτυχία μόνο εάν υπάρχουν αν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ε, μέσα από τον οποίο θα εφαρμοστούν. Τώρα, η συμπερίληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στις συνάψεις των συμβάσεων. Όντω ε, θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και εδώ θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτή οι αναθέτουσες αρχές να έχουν την ευκαιρία να κατανέμουν την, συμβάσει συμβάσεις σε ε, μερίδια, αν θέλετε, σε παρτίδες και η κατανομή σε παρτίδες ε, είναι μια πόρτα εισόδου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όταν δεν υπάρχει αυτού, δεν υπάρχουν αυτές οι παρτίδες, πάλι υπάρχει μια ε, διαδικασία ανάθεσης σε υπεργολάβους. Άρα και μέσω αυτού του έμεσου τρόπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συμμετέχουν στις ε, δημόσιες συμβάσεις. Άρα εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στις δημόσιες αρχές και στις ανατέψεις αρχές για την σύναψη των συμβάσεων. Τώρα, είμαι στη διάθεσή σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζή Μαρικάκη, τον κύριο Χέγγελ, τον κύριο Κρόιτσμαν, την κυρία Ρούλε, τον κύριο Αρμπούρ, τον κύριο Ντε και τον κύριο Σαλβίνη, τον κύριο Σαλβίνη, τον οποίο δεν γνωρίζω γιατί δεν τον είδα σε καμία συνεδρίαση. Α, τι ωραία, εδώ είναι. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνωρίζω. Λοιπόν, ε, γίνανε πολλά, πολλές ε, συζητήσεις ε, με τους σκιώδεις συγητές και θα υπάρξουν και άλλες, διότι είναι και αμφιλογόμενο λίγο το θέμα. Υπάρχουν πολλές ιδέες διαφορετικές και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε δύο οδηγίες και που θα εισάγουν ε, ε, βελτιώσεις ε, και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις αναθέτουσες αρχές που ακόμα, όπως και οι δικοί μου, προσπαθούν να χωνέψουν τις οδηγίες του 2004 και ακόμα δεν είναι έτοιμες. Επομένως, χρειάζεται μια πλούστευση των διαδικασιών, πιστεύω. Σας ευχαριστώ και σας ναι. ακούω με ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε για την εισαγωγή σας. Πρωτού προχωρήσουμε. Να σας ζητήσω απλά, επειδή όσοι έχουν εξοικειωθεί γνωρίζουν τι είναι τα κλάστερς, οι κατηγορίες, κατηγοριοποίησεις, αλλά από τους εκτός ιστάμενους και μη εξοικειωμένους θα μπορούσατε να συνοψίσετε τι συμφωνήσαμε στη διαδικασία εργασίας και δεν γνωρίζω κατά πόσο έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ότι έχουμε 1593 τροπολογίες όλες που αφορούν αυτές τις πτυχές που συζητούσαμε. Και έχουμε και πολλά, πολλούς ευρωβουλευτές που θα ήθελαν να συνεισφέρουν με κάποια αρχικά σχόλια εγκάρσια για όλες τις τροπολογίες. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αυτά λοιπόν. Και είχαμε και ένα χρήσιμο έγγραφο εργασίας για το κλάστερ που θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη μετά τη συνεδρίαση ώστε όλα τα μέλη οι ευρωβουλευτές να γνωρίσουν πώς τα προσεγγίζουμε όλα αυτά, διότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις. Μπορείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αποσαφηνίσετε κάποια πράγματα και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να δραχθώ τη ευκαιρία να καλωσορίσω τον Κλάους Βίνερ και τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς θα έχουμε ευκαιρία να ακούσουμε κάποιες παρατηρήσεις για τις τροπολογίες στη συνέχεια. Τώρα Μακ Ταραμπέλα μπορείς να μας πεις πώς έχουν αυτά τα πράγματα προτού περάσουμε στις επόμενες φάσεις για την εξέταση αυτών των τροπολογιών. Θα ήταν επικοδομητικό ευχαριστώ. Οι κλώστερ τώρα ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα της Προεδρίας της Δανίας να γίνει ένας χωρισμός της οδηγίας θεματικά που έχει συγκεκριμένα άρθρα. Έγιναν 10 κλώστερ, ανέφερα τις 5 πρώτες για καλύτερη επιλογή της διαδικασίας. Μετά έχουμε τη στρατηγική για τις δημόσιες ε, συμβάσεις. Μετά το θέμα που έχουν να κάνουν με, με τις ε, προσφορές. Στην 7 έχουμε την πρόσβαση στις, των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες προσφορές. Η έκτη ε, και μετά οι έβδομοι έχουν να κάνουμε με τις ε, για, θέματα που έχουν να κάνουν με τις προθεσμίες βασικά. Μετά έχουμε, ε, έχουμε μετά τη διαδικασία η οποία λέγεται υγιής διαδικασία ε, επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν προσφορές οι οποίες δεν είναι πολύ χαμηλές κτλ. Μετά έχουμε το θέμα της καλύτερης διακυβέρνηση με μια διαδικασία ενημέρωσης. Μετά έχουμε την περίπτωση όπου έχει να κάνει με το πεδίο εφαρμογής, εφαρμογής ε, θέματα πλαφών και θέματα ονοματολογίας και ορισμού. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ε, για να υπάρχει καλύτερη σαφήνεια έχουμε δύο οδηγίε οι οποίε ενώθηκαν και έχουμε τον μεγάλο αριθμό των τροπολιών που αναφέρατε. 13 είχαμε στο Στρασβούργο την τελεσμένη εβδομάδα μια συνάντηση. Σήμερα έχουμε τη, τη ε, συζήτηση αυτή. Επίσης θα έχουμε μια δεύτερη συζήτηση 5 Νοεμβρίου για το cluster 6 μέχρι 10 και μετά στη συνέχεια θα έχουμε το shadow meeting 20 ε, ε, Σεπτεμβρίου. 25 Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια συνάντηση για την κλώστερ 3, 7, 8. 10 Οκτωβρίου τώρα θα έχουμε συζήτηση για το κλώστερ 2 που είναι εμβληματική θα λέγαμε περίπτωση. 18 Οκτωβρίου shadow meeting για να κλείσουμε την Cluster 2 και να ξεκινήσουμε τη 10. 25 Οκτωβρίου Cluster 10 θα έχει τελειώσει και ενδεχομένω η 9. 7 και 13 Νοεμβρίου τώρα κανονικά ένα shadow meeting για την 5η και 6η Cluster και τέλη Νοεμβρίου και ελπίζουμε να είναι η τελευταία συνάντηση ένα shadow meeting για τα τελευταία προβλήματα που θα πρέπει να διασαφινιστούν. Και 28 Νοεμβρίου συζήτηση για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. 29 Νοεμβρίου επαναλαμβάνω, στη συνάντηση ΙΜΚΟ, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ε, ε, αυτά έχουν προβλεφθεί. Θα δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτή τη διαδικασία. 29 Νοεμβρίου επαναλαμβάνω, στη ΙΜΚΟ. 10 Δεκεμβρίου προβλέπεται η ψηφοφορία ε, τμηματικά για την οδηγία, μάλλον ή 10 Δεκεμβρίου στο Δεκέμβριο ή 18 Δεκεμβρίου εδώ πριν τα Χριστούγεννα, για να κλείσουμε αυτές τις δύο οδηγίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια επιθυμία από τον Φρανκ Ένκελ, αλλά νομίζω οι περισσότεροι έχουμε αυτό τον, αυτή την επιθυμία. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ήταν χρήσιμο αυτό για να γνωρίζουν όλοι περί τίνο πρόκειται και για τους συντονιστές που το απόγευμα θα συντονιστούν και θα συναντηθούν για να ε, συζητήσουν και εξετάσουν το χρονοδιάγραμμα που είναι και ευθύνη τους. Αλλά νομίζω πιστικά παρουσιάσατε τα πράγματα και έχουμε και τις υποδομές για να υποστηριχθεί αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει να δημοσιευθούν αυτά ευρύτερα, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν περί πρόκειται, να εξοικειωθούν και να ξέρουν πώς προχωρούν οι συζητήσει. Ο Κλάου Βινέρ θα θέλει και αυτός να συνεισφέρει, πιστεύω, επίση από πλευρά του. Στη συνέχεια, λοιπόν, τώρα θα ήθελα να έχουμε απαντήσεις, ε, παρεμβάσεις απαντήσεις από τους σκιώδεις εισηγητές και από άλλους ευρωβουλευτές που θα ήθελαν να συζητήσουν κάποιες πτυχές. Η κυρία Στάιλερ έχει ήδη πει θέλει να παρέμβει, είναι η πρώτη. Γκέπαρτ και Ζουβά είναι επίσης στον κατάλογο. Γκέπαρτ, Ζουβά, Στάιλερ, άλλοι που θα ήθελαν να παρέμβουν. Και ο κύριος Σβάμπ, εντάξει. Ας ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις λοιπόν. Έγκελ και μετά Χατζημαρκάκης. Κύριε Έγκερ, έχετε τον λόγο λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή να ευχαριστήσω για αυτήν την πρώτη, τον πρώτο γύρο. Βλέποντας την προσέγγιση τη δική του, πολύ πιο αριθμητική και μαθηματική θα έλεγα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτό το τομέα πραγματικά έχω δύο οι οποίες δεν μου λένε τίποτα. Εγώ έχω μια προσέγγιση πιο λυρική, όπου η διατύπωση των πραγμάτων γίνεται με έναν τρόπο, σε οποιαδήποτε ε, γλώσσα φυσικά, αλλά με ένα πιο λυρικό τρόπο. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό με τους αριθμούς που μας έδωσε ο Μάρκα, ο οποίος έχει δίκιο από την πλευρά του φυσικά. Ε, εγώ επίσης δεν κρύβω το γεγονό ότι ε, βλέποντα ε, όλο αυτό το κείμενο και ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση απόψεων η οποία έχει να κάνει με τις πολιτικές ομάδες. Έχει μια προσέγγιση εδώ πέρα η οποία καλύπτει γενικά το, το ΕΛΚ φυσικά. Οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν προσωπικές απόψεις διαφορετικές. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Θα ξεκίνησω λέγοντας η νομοθεσία για τις δημόσιες ε, προσφορές δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Αυτό είναι εκεί μου απόψη. Το έχω δει και με δύο εκθέσεις πρωτοβουλία που είχαμε κάνει στην αρχή αυτής της ε, θητείας. Υπάρχει στρατηγική άποψη. Όμως δεν μπορεί νομοθετικά να καλύψει τα πάντα για τις δημόσιες προσφορές. Αυτή είναι η άποψη της πολιτικής μου ομάδας. Και αυτό ισχύει και εδώ. Δεν θα είμαστε σε θέση δυστυχώς να βελτιώσουμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με θετικούς τρόπους. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και είναι σαφές για μας ότι για αυτή τη στρατηγική προσέγγιση Υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Είναι κριτήρια τα οποία τα προφέρουν μη. Αυτό δημιουργεί μια, κάποιον να σκεφτεί το κρέας. Εγώ θα τιμήσω τη λέξη μα και να επιλέξουμε τις πιο προνομιακές προσφορές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να συγκεντρωθούμε πιο προσεκτικά και να κοιτάξουμε να επιλέξουμε τις πιο οικονομικές επιλογές σε σχέση με το γενικότερο κλίμα. Αυτό Άρα η προσέγγιση που να κάνουμε είναι για, που έχει να κάνει με τις τιμές τις πιο χαμηλές. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη. ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από την αρχή ότι θα υπάρξουν κάποιες αποκλήσεις ανάμεσα, ανάμεσα μας και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Ε, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και στη δική μου ομάδα επίσης όπου υπάρχει η θέληση να μειώσουμε τα, το κόστος μεταφορών για να βοηθήσουμε ε, τοπικά την οικονομία. Εγώ προσωπικά θεωρώ αντιθέτως ότι υπάρχει μια δυνατότητα να επιμείνουμε στην παραγωγή κάποιου θέματος ή να κοιτάξουμε τα θέματα υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε μια θα λέγαμε κοινοτική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό κατά με είναι ίσως δυνατό, αλλά δεν βλέπω τη σημασία να δώσουμε πολύ έμφαση σε κάτι που έχει τοπικό, περιφερειακό χαρακτήρα. Υπάρχει επίσης το θέμα της αμοιβαιότητα. Τι γίνεται εδώ τώρα. Εδώ πέρα συνδέεται και με ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν νομοθετικά μέσα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε και να μην τα συγχαίουμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία μπορούμε να τάξουμε στην νομοθεσία την οποία προβλέπουμε τώρα για τις δημόσιες προσφορές. Εγώ θα ήθελα να είμαι σαφής. Επιλέγω την πρώτη επιλογή και όχι τη δεύτερη. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά την νομοθεσία που έχει να κάνει με τι δημόσιε προσφορέ και φυσικά να προκαταλάβουμε και τι συνέπειε που μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον. Να μην προσπαθούμε να προσεγγίσουμε θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν πρόκειται στο μέλλον να επαληθευτούν. Τώρα, για την εταιρική σχέση, για το διάλογο και την ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα να πω ότι όλοι η οδηγία θα πρέπει συνολικά να περάσει σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει συνολικά η οδηγία να ενσωματωθεί. Δεν πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, μια α ή β χώρα να προσπαθήσει να κάνει κάποια επιλογή, να μην υιοθετήσει, εγκρίνει, συγγνώμη, συνολικά την οδηγία. τώρα για κάποιες ε, παραλλαγές που μπορεί να υπάρχουν, αν παίζει ρόλο αυτό, αν συμβάλλει στην ε, καινοτομία, καλώς. Το, η βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ πέρα ε, ανέφερε πολλά ο Μάρκ. Για την κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία. Εδώ έχουμε μετά πνευματικά δικαιώματα και τι ακριβώς πρέπει να πράξουμε. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε μια ειδική νομοθεσία. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα στην πράξη, στη σύλληψη και στη νομική πτυχή. Αν έχουμε μια ειδική νομοθεσία, δημιουργεί κανείς, ευρίσκει κανείς νέες έννοιες για να μπορέσει να κάνει μια εφαρμογή. Δεν υπάρχει αυτό το κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία παραγωγής είναι κάτι που εφήβρε ο Μάρκ. Εγώ θα έχω κάποια προβλήματα με αυτό. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε με αυτή την έννοια. Πού θα καταλήξει ακριβώς. Τώρα, σε κάτι άλλο. Την πρόσβαση το, για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μας ε, αφορά σήμερα το πρωί για τις ε, δημόσιες προσφορές. Συμβάσεις, συγγνώμη. Να πω κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση όταν γίνεται συνολικά ένας καταμερισμός, ένας χωρισμός, Τι θα γίνει δηλαδή, θα δημιουργήσουμε τώρα μια αρχή εν ονόματι του συνόλου να ε, εγκαταλείψουμε τομεακά διάφορους χώρους. Υπάρχει το κριτήριο ότι το βασικό κριτήριο, να έχουμε κάποιο κατόφλι όχι. Θα υπάρξουν συμπληρωματικά προβλήματα, τα οποία θα είναι δύσκολα να λυθούν. Και δεν οδηγούμαστε σε κάποια απλοποίηση όπως επιθυμούμε. Το να πει κανείς, το να προσπαθεί κανείς να προσδιορίσει πώς ακριβώς γενικότερα ή ειδικότερα θα λύσει ένα θέμα, Όλα αυτά θα πρέπει να τα λύσουμε, να μην τα περδέψουμε τα πράγματα και θα το δούμε όταν φτάσουμε στις ε, λεπτομέρειες. Κάτι που με ανησύχησε στην αρχή έχει να κάνει με το θέμα του κατοφλιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεθνείς ε, δεσμεύσεις. Δεν είναι εύκολο και λογικό να αλλάξει κανείς κάποια κατόφλια. Εγώ θα κάνω μια πρόταση στους συναδέλφους. Με αυτούς που συνεργάζομαστε συγκεκριμένα. Να δούμε μια μεταβατική περίπτωση να δούμε όταν θα ξαναγίνουν διαπραγματεύσεις με τις, σε διεθνές επίπεδο να κοιτάξουμε, να δούμε αυτά τα θέματα ούτως ώστε τα θέματα επίπεδου κατοφλού να είναι πιο ρεαλιστικά. Και τώρα για τις υπεργολαβίες. Στο μέλλον, κατεμέ να είμαστε ξεκάθαροι τι ακριβώς κάνουμε με τις επροβολαβίες, ποιο ακριβώς αναλαμβάνει κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχει το θέμα να υπάρχει μια διαφάνεια στην αλυσίδα υπεργολαβιών, να, γίνει, να καθοριστούν αυτές οι διαδικασίε, να γίνεται μια αξιολόγηση από την αρχή, ποιο είναι αυτό ο οποίο θα παρέμβει στη διαδικασία υπεργολαβίας, με ποιο τρόπο, για ποιο όγκο παραγωγής να γίνει ένα τέτοιο λόγο και να ξέρουμε ότι στο τέλο αυτό που αναλαμβάνει την υπεργολαβία είναι ικανό να διεκπαιρεώσει κάτι. Ε, πάει πολύ μακριά αυτό το θέμα ότι οποιαδήποτε επιχείρηση Φερπίν θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία των υπεργολαβιών. Και είναι αδύνατο κατ' εμέ να περιορίσουμε τον αριθμό αυτών οι οποίοι ε, λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις προκαλαβίες θα είναι αυθαίρετος ο τρόπος ε, ορισμού. Ποιο ποσοστό θα καθοριστεί κτλ. Δεν μπορεί κανένα να ελέγξει τον α, β αριθμό. Θα πρέπει φυσικά να είναι σαφές ότι όλοι θα πρέπει να ξέρουν τι κάνει ο καθένας, αλλά να αποφύγουμε τις υπερβολές πράγματα τα οποία πραγματικά δεν φταίχουν ουσιαστικά. Φυσικά να δούμε και με ένα ορθό και λογικό τρόπο για θέματα που έχουν να κάνουν με, την, με τις Αυτά σε γενικές γραμμές σαν πρώτη προσέγγιση κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώντας φυσικά τον συνάδελφο Μάρκ Ταραμπελά για το έργο του σε μια δύσκολη περίοδο. Και τέλος να πω ότι χαίρομαι ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί. Ευχαριστώ. Um, thank you very much, Mr. Um, for the Group. Σα ευχαριστούμε εσεί για την ομάδα τη Άλντε, κύριε Χατζημαρκάκη. Θα ήθελα να εκθέσω την θέση τη Άλντε Κανονικά ο Γιούργεν Κρόισμαν θα το έκανε, αλλά έχει υποχρέωση σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Και γι' αυτό ανακατηγορία κλάστερ θα τα εξετάσω ώστε να παρουσιαστεί και το αποτέλεσμα των εσωτερικών μας διαβουλεύσεων εχθέ και να σας τις ανακοινώσω για την κατηγορία 1 για την επιλογή και τα τα κράτη-μέλη στις ε, δημόσιες αρχές θα έχουν τις ίδιες αρχές που θα ισχύουν. Αυτή είναι η θέση μας. Σε νέε διεργασίες θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτόματα θα είναι διαφανεί και δίκαιες αυτές οι διεργασίες. Αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζεται αυτό. Θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρχει περιθώριο για διαφθορά και νεποτισμό <clears throat> η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να είναι πιο σύντομη από ό,τι μέχρι σήμερα, αλλά πιο μεγάλη από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μια μέση οδό για συμβιβασμό για την κατηγορία 2, στρατηγική χρήση των δημόσιων προμηθειών και προσφορών. Αυτή το δυνατόν λιγότερες, περιορισμού περιορισμούς θα πρέπει να έχει, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια επίσης, απαιτούμε αυτή είναι η θέση μας, για τι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι δυνατόν στις συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής να αναφερόμαστε, όσον αφορά την ε, αναλογικότητα σε σχέση με τις ε, εντολές. Ε, οι δημόσιες αυτές προσφορές θα πρέπει είτε να επιλέγουν το πιο οικονομικό, την πιο οικονομική προδιαγραφή ή την χαμηλότερη τιμή να εφαρμόζουν για την επιλογή. Για τον καθορισμό του, της πιο ευνοϊκής προσφοράς θα πρέπει <clears throat> αυτοί που θα αποφασίζουν να μην αναφέρονται μόνο σε κοινωνικά στοιχεία τα οποία θα ξεπερνούν τα νομικά πλαίσια αυτό είναι ένα σημείο βέβαια το οποίο γνωρίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε σε βάθος και που το βλέπει διαφορετικά κάπω ο εισηγητή. Για την καλή συνεργασία η Άλντα ευχαριστεί φυσικά και είναι αυτονόητε αυτέ οι ευχαριστίες Καθορισμό αυτών των ε, διεργασιών πρέπει να ε, επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σχέση με το αντικείμενο αυτών των ε, διεργασιών και θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωστοποιούνται οι προσφορές αυτές ε, πριν από την λήψη απόφασης. Ε, περνάω στην κατηγορία 3 όσον αφορά τα τεκμήρια απόδειξης. Χαιρετίζουμε την εισαγωγή ενός πάσου, ενός διαβατηρίου δεν θα πρέπει να απαιτούνται περαιτέρω ε, στοιχεία τα οποία δεν θα εμπεριέχονται σε αυτό το πάσο, σε αυτό το διαβατήριο. Αυτό το διαβατήριο όμω θα μπορούσε να εμπεριέχει περαιτέρω στοιχεία που θα αφορούν του ε, οικονομικά εμπλεκόμενου. Για την κατηγορία 4, κλάστε 4, ηλεκτρονικές εντολές ε, και καταχωρήσεις. Θα πρέπει από κοινού με τον Μάκομ Χάρμπορ εδώ να δούμε το τι προτείνουμε προτείνουμε μια κλιμακούμενη προθεσμία. Μέχρι την 1η Πρώτου 2017 τα κράτη-μέλη θα πρέπει τουλάχιστον 70% των ε, ε, εντολών αυτών ηλεκτρονικά να τις ε, διευθετούν. Μέχρι το 2020 θα πρέπει 100% να έχουμε καταφέρει να γίνονται όλα αυτά ηλεκτρονικά. Βλέπω συγκατανεύει ο Πρόεδρος. Αυτές σε δύο κλίμακες διεργασίες φαίνεται για μας ότι είναι πιο λογικές και έχουν μεγαλύτερο νόημα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει διαφορετικές ημερομηνίες. Τελευταία κατηγορία, πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να υποχρεώνονται να ε, εξετάζουν ε, τις ε, πληροφορίες αυτές ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να υποφεληθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ώστε μέσα στη γνωστοποίηση των εντολών σε σχέση με τις προσφορές να αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπεργολαβίες και την έγκρισή τους, όπου στοιχεία για αυτές τις ε, υπεργολαβίες, θα, μπορούν να, θα μπορούν να απαιτούνται και να γνωστοποιούνται. Σε σχέση με τους ε, ιδιώτες ε, και τις υπεργολαβίες θα πρέπει σε ένα εθνικό πλαίσιο αυτό να είναι εφικτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτική προδιαγραφή για πανευρωπαϊκό τέτοιο πλαίσιο. Αυτή είναι η θέση της ομάδας μας. Ευχαριστώ τον Μάκ Ταραμπέλα για την πολύ καλή συνεργασία μας. Thank you, Ευχαριστούμε κύριε Χατζημαρκάκη, κυρία Ρούιλε. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να προσθέσω τι ευχαριστίε μου προ τον εισηγητή. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ωστόσο, και απευθύνω έκκληση σε όλου του ευρωβουλευτέ που είναι στην αίθουσα, ωστόσο, επαναλαμβάνω, θα είναι δύσκολο το εγχείρημα. Αυτό που θέτει ο εισηγητή στο επίκεντρο των όσων εξήγησε. Η απλούστευση δηλαδή των δημόσιων αυτών προμηθειών και αγορών. Αν δει κανεί τον τεράστιο αριθμό τροπολογιών και αν δει κανεί πόσο παρεκκλίνουν οι διαφορετικέ θέσει και προτάσει μεταξύ του σε σχέση με αυτέ τι τροπολογίε πεδίο εφαρμογή, όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι σημαντικέ οι έννοιε αυτέ και για την απλούστευση. Έτσι ξεκινήσαμε τη δουλειά. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τέτοιου είδου συμβάσει που βρίσκονται πάνω από το κατόφλι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελέτη τη τόνισε για άλλη μια φορά ότι μόνο τα επιπρόσθετα γραφειοκρατικά βάρη θα είναι 30, ε, ε, ε, είναι ένα τεράστιο ποσό και σε σχέση με τις διαβουλεύσεις μας φτάνουν πολλές φορές στο 1 τρίτο της συνολικής αξίας. Αυτό είναι υπερβολικό. Θέλουμε όλα αυτά να τα απλουστεύσουμε και να δημιουργηθεί μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Μόνο τότε όμως θα τα καταφέρουμε όλα αυτά αν περιορίσουμε το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή να πούμε ότι οι δημόσιες προμήθειες και θα πρέπει να διαμορφώνονται σε ένα διαφανές πλαίσιο. Να μην υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος κανενός. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ως υποκατάστατο κάποιους κανόνες και κανονισμούς που θα υιοθετήσουμε σε αυτό το πλαίσιο και που δεν συσχετίζονται άμεσα με αυτές τις προμήθειες. Αυτό έχει τη σημασία του, διότι αν όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να πορευτούμε προς την κατεύθυνση της πιο ευνοϊκής προσφοράς που θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο ή να είναι η μόνη προσφορά που θα μπορεί να εγκρίνεται, μόνο τότε θα μπορούμε να τα πετύχουμε στην τελική εφαρμογή αν βελτιώσουμε τα πράγματα για την νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Ξέρω την πρακτική ε, πώς ακολουθείτε σήμερα υπάρχει ο φόβος ότι στη μία ή άλλη περίπτωση, στη μία ή άλλη περίπτωση σε εισαγωγικά οι τιμένοι, εκείνοι που δεν ευνοήθηκαν σε σχέση με την τελική επιλογή, θα προσφύγουν σε δικαστήρια. Γι' αυτό με αυτή την οδηγία δεν πρέπει να δημιουργηθεί νομική αβεβαιότητα ή ανασφάλεια. Πρέπει να βελτιωθεί το αντίθετο ακριβώ. Πρέπει να συμβεί να βελτιωθεί η νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Τώρα, κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν προβλήματα. Αφενό οι προσδιορισμοί, οι ορισμοί. Εξαιρετικό ακούγεται να έχουμε ορισμού για την κοινωνική αηφορία όσον αφορά αυτέ τι εντολέ. Αν τώρα εισαγάγουμε όμω κάποιε νέε έννοιε που δεν τι προσδιορίζουμε επακριβώ και δημιουργείται ασάφεια, τότε μεριμνούμε φυσικά ώστε η νομική αβεβαιότητα πάλι να αυξηθεί και όχι να μειωθεί. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να εξετάσουμε ακριβώ πώ θα μπορέσουμε το στόχο μα να τον πετύχουμε. Για τι ε, δημόσιε αρχέ να είναι όλα αυτά εφικτά και να μπορούν να λειτουργήσουν και να αυξηθεί η νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό σε, όλες, ε, σε όλα τα πλαίσια αυτά να διασφαλιστεί η νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Τώρα, για τη διαφάνεια και ισότητα μεταχείρισης. Όσοι είναι υπέρ αυτών των ενιών πρέπει να μεριμνήσουν οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την εκτέλεση των εντολών πάντα να έχουν ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τον τελικό στόχο αυτού του εγχειρήματο. Γιατί διαφορετικά μπορεί αυτή η διαφάνεια να διακυβεύει την ε, ε, αποτελεσματικότητα. Ένα άλλο σημείο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο είναι σημαντικό για μένα και για το οποίο σήμερα συζητήσαμε ευρέω. το θέμα των υπεργολαβιών και των υπεργολάβων είναι φυσικά ευκταίο να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτό το πλαίσιο. Όμως, οι υπεργολάβοι και οι υπεργολαβικέ επιχειρήσεις δεν είναι μόνο στον τομέα των οικοδομών ή στον τομέα των, κοινωνικών θεμάτων ή στι γενικότερες υπηρεσίες. Είναι ένα γενικότερο θέμα. Αν περιορίσουμε τον αριθμό των υπεργολάβων, θέλω να ξέρω Πώς είναι δυνατόν να αγοράσει κάποια δημόσια αρχή να προμηθευτεί ένα όχημα για την πυρόσβεση. Γιατί κάθε όχημα το οποίο αγοράζεται ε, προβλέπει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα για αυτή την προσφορά ή για αγορά ηλεκτρονικών εγκεφάλων. Πώς θα γίνουν αγορές ηλεκτρονικών εγκεφάλων όταν περιορίζονται οι υπεργολάβοι σε τρεις αποκλειστικά και μόνο. Θα είναι ανέφικτο, θα είναι, δεν θα είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε και μεγάλη αλυσίδα ε, στοιχείων ανταλλακτικών. Πρέπει όλη την αλυσίδα να την εξετάσουμε. Φυσικά έχω προβλήματα για το τι γίνεται στον οικοδομικό τομέα αυτή τη στιγμή. Αν έχουμε όμως κάποιες ε, προδιαγραφές που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν εξυπηρετούμε κανένα. Θέλω να περάσω σε ένα σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Τις δημόσιες αυτές εντολές δεν θα πρέπει να τις επιβαρύνουμε με περαιτέρω όρους και προδιαγραφές που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πολλέ φορέ είναι μικροϊπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν σε αυτά τα πλαίσια. Τώρα, να ελέγξουν όλους τους παρόχους ε, και ε, όλους τους εμπλεκόμενους, ε, αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας και των τελωνίων. Οι μικρο... Και δεν μπορούν να τα καταφέρουν αυτοί πάλι. Πρέπει να είμαστε αναλογικοί, να τηρήσουμε την αρχή της αναλογικότητας, να μην υπερβάλλουμε με άλλα λόγια σε σχέση με την διεύρυνση των πλαισίων. Η άποψή μου είναι ότι πολλές ε, πολλές υπηρεσίες, δήμοι, κοινότητες έχουν ιδιαίτερο συμφέρον οι συμβάσεις αυτές με οικολογικές, κοινωνικές και ηθικές αρχές ε, να διευθετούνται. Αλλά αν δεν υπάρχει ασφάλεια, νομική βεβαιότητα και υπάρχουν περιορισμοί, θα ακολουθούν την πιο απλή ε, οδό και αυτή θα είναι η πιο ευνοϊκή προσφορά. Ευχαριστώ. Uh, thank you uh, uh, ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρούιλε. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σύντομα σχόλια εξ ονόματος της ομάδας μου. Διότι έχουμε καταθέσει και εγώ και ο συνάδελφος κάποιες τροπολογίες, αλλά όλες διασυνδέονται και θα πρέπει να δούμε τα κύρια θέματα για τα οποία συζητούμε εδώ σήμερα και σε αυτά να επικεντρωθούμε. Κατανοώ και παρακολουθώ αυτά τα οποία είπε με σαφήνεια η κυρία Ρούλε. Πρέπει οι διαδικασίες αυτές θέλουμε να ξεκινήσουν αυτές οι διαργασίες και να ενθαρρυνθούν οι καλύτερες πρακτικές για αυτές τις προμήθειες και αγορές. Έχουμε περιορισμούς ε, αυτή τη στιγμή και επιβαρύνσεις που δεν επιτρέπουν στους πολίτες ε, και πελάτες να επιλέξουν την καλύτερη λύση για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ιδιαίτερα όταν έχουμε και πτυχές ε, όπως την κοστολόγηση που βλέπουμε ότι αποτελεί όλο και περισσότερο στοιχείο το οποίο εξετάζεται πρέπει να έχουμε σαφές, κατευθυντήριε γραμμές πώ θα διαμορφώνονται όλα αυτά και άλλα στοιχεία τα οποία θα συνεισφέρουν ώστε να μπορεί ο εκείνος που προσφέρει την πιο ευνοϊκή προσφορά να μπορεί να επιλέγει. Έχουμε κάποιες διαφωνίε, βέβαια για το τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτούς τους ορισμούς. Όμως πιστεύω ότι αν έχουμε, αν περιοριστούμε στις οικονομικά πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, αυτό θα φωτίσει την πορεία και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. δεύτερη πτυχή αφορά το συνολικό θέμα των διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Ουσιαστικά οι διεργασίες αυτές να μπορέσουν να καταστούν καλύτερα προσαρμόσιμες και προσαρμοστές στις ανάγκες των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη να ε, κάνουν τέτοιες ε, αγορές ε, και και προμήθειες. Όμως η διαφάνεια όλων των διεργασιών σε σχέση με τον ανταγωνισμό για την υποστήριξη, για την ενθάρρυνση ε, των επιχειρήσεων που θα μπορούν να ε, προσέρχονται και να υποβάλουν προσφορές σε σχέση με πελάτες που θα μπορούν να ικανοποιηθούν από αυτές τις προσφορές, διατηρώντας δηλαδή τα στοιχεία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, αλλά έχοντας τελικά πιο προσιτές τιμές και πιο αποτελεσματική διεργασία για αυτές τις τιμές. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε και όχι να έχουμε ένα ακριβό πλαίσιο πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούμε. Δεν πρέπει να υπάρχει νομική αβεβαιότητα, δεν πρέπει να υπάρχουν ε, πολλές ε, ε, δυνατότητες υπεκφυγής και να μην μπορεί κανείς να κατανοήσει στο πού βρίσκεται σε όλα αυτά. Συνδέεται με αυτό και όπως όλοι γνωρίζετε το ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ήταν προπομπός, ήταν πρωτοπόρο στο επιχείρημα να υπάρξει μια διαδικασία προμηθειών ώστε να ενθαρρυνθούν οι πιο καινοτόμε λύσεις. Προκλήσεις για εκείνου που θα υποβάλουν τέτοιες προτάσεις για προσφορέ. Ε, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο τέλος τέλος ε, με τα όσα προτείνονται και προσφέρονται. <clears throat> Νομίζω είναι πολύ επενέσιμη αυτή η προσπάθεια λοιπόν. Κάναμε κάποιες προτάσεις. Νομίζω πρέπει να βελτιωθούν αυτά τα πλαίσια. Είναι ένα νέο ε, πεδίο αυτό στο οποίο κινούμαστε και θα δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει πρόκληση για τη δική μα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτά ζητήσαμε να γίνουν και πρέπει να συνεργαστούμε να βελτιωθούν στο μέγιστο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική προσέγγιση που υιοθετήθηκε και το επικοδομητικό πλέγμα σε σχέση με τι διαβουλεύσει. Πολλέ τροπολογίε βρίσκονται στο τραπέζι, συνάδελφοι, αλλά πολλέ από αυτέ στοχεύουν στην ίδια κατεύθυνση. Να υπάρχουν βελτιώσει ε, στι Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες σε αυτό το πλαίσιο για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση και το ίδιο το Συμβούλιο παράλληλα εργάζεται πρέπει να πω και γύρω από αυτές τις συζητήσεις με τον ίδιο τρόπο τοποθετείται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό εξίσου και κάποιες άλλες παρατηρήσεις τώρα ο κύριος Κατζημαρκάκης νομίζω ανέφερε τις τροπολογίες μας για την ηλεκτρονική, τις ηλεκτρονικές δεν μειώνεται με κανένα τρόπο η σπουδαιότητα των ηλεκτρονικών προμηθειών. Πρέπει να δουλέψουμε παράλληλα με τις προσπάθειες των κρατών μελών και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα. Έχει κέρια σημασία αυτό. Κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν σήμερα, αλλά πρέπει να αναφερθούν σε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων είναι το ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι υπάρχει ανάγκη για τα κράτη-μέλη να βελτιωθεί η συνολική ε, παρακολούθηση αυτών των διεργασιών. Όχι όμως ισοπεδωτικά με μια πρόταση που θα ρυθμίζει τα πάντα. Δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να μειωθεί η σπουδαιότητα τη συμμόρφωσης με του κανονισμού και του κανόνε. Πολλέ τέτοιε συμβάσει πρέπει να μπορούν να εντάσσονται μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα δημόσιων προμηθειών και αγορών, αλλά όχι ισοπεδωτικά, υποχρεωτικά. Και παρόμοια, βελτιώνοντας τις διεργασίες και διαδικασίες, νομίζω η αυξανόμενη χρήση των δηλώσεων που υποβάλλονται από τους ε, ίδιους τους ε, εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενου, είναι σημαντική υπόθεση. Και ενώ και το Ευρωπαϊκό διαβατήριο είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Οι αυτοδηλώσεις μπορούν να, να συνεισφέρουν ε, όσον αφορά την, το συνολικότερο πλαίσιο, όχι όμως να επιβαρύνουν γραφειοκρατικά. Να δούμε αν θέλουμε στο τέλος τέλος να ε, καταλήξουμε σε κάποιες τέτοιες λύσεις. Και για την πρόσβαση ως άξονα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικό για τις αρχές και τους πελάτες να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εξετάσουν εξετάζουν τα θέματα των ΜΜΕ. Πρέπει όμω να μην έχουμε υπερβολικά περιοριστικά πλαίσια με υπερβολικά πολλέ προδιαγραφέ και κανονισμού. Θα πρέπει να εξετάζετε εκάστοτε τι είναι το καλύτερο για τον καθένα. Αλλά πάντα να λαμβάνονται και οι ανάγκε των ΜΜΕ. Να υιοθετούνται διεργασίε ώστε να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, σε δυσμενέστερη θέση ΜΜΕ. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε σφαιρικά αυτέ τι διεργασίε. Προσβλέπουμε στο να εξεταστούν οι τροπολογίε από του συναδέλφους και του σκιώδη οι κατά τους επόμενους μήνες ε, με το πιο αποτελεσματικό τρόπο για να καταλήξουμε σε σημαντικές ε, και λογικές βελτιώσεις. Νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν λίγοι τομεί στους οποίους έχουμε ριζικές διαφωνίες και εκεί πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα. Κατά τα άλλα έχουμε νομίζω κοινέ απόψεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Κάποιες πτυχές για την απλούστευση αυτών των διεργασιών το τμήμα Α, τμήμα Β, part A, part B για αυτές τις υπηρεσίες και το θέμα της απλούστευσης και για η προσπελασιμότητα για κάποιες υπηρεσίες πρέπει να εξετάσουμε κάποια πράγματα και να δούμε τι μπορεί να γίνει, να υποβληθούν και κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες. Προσβλέπουμε λοιπόν στο να συνεργαστούμε με τον εισηγητή προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, ο κύριο Σαλβίνη είναι ο τελευταίο από του κοιόδη εισηγητέ. Θέλετε να παρέμβετε σε αυτή τη φάση, κύριε Σαλβίνη. Α, ο κύριο Ντε παρακαλώ, συγγνώμη. Ο κύριο Ντε Κύριο Ντε πρώτα, μετά ο κύριο Σαλβίνη. Και μετά θα ξεκινήσουμε με του πέντε εναπομείναντε ομιλητέ. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να πω πώς ακριβώς ε, αντιμετωπίζει το θέμα η ομάδα μου. Έχουμε χάσει τις, ε, την πρώτη συνάντηση εξαιτίας των εκλογών που είχαμε στις κάτω χώρες. Σε σχέση με αυτά που είπε τώρα η κυρία Ρουλ, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ, δηλαδή χρειάζεται ένα, ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι απλουστευμένο και καλύπτεται νομικά. Όταν βλέπει κανείς πως έχει εξέλιξη, ε, καταλήγουμε σε ένα προϊόν το οποίο μάλλον θα λέγαμε είναι πιο περίπλοκο. Εγώ τώρα σκεφτόμουν με την πρώτη κατηγορία, Closer, οι δημόσιες συμβάσεις ε, πρέπει να παίζουν ένα στρατηγικό ρόλο, να υπάρχει διαφάνεια και οπωσδήποτε οι, οι, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να συμβάλλουν στο να υπάρξει μια πολιτική η οποία καλύπτει πτυχές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αυτό πρέπει να περάσει μέχρι το επίπεδο των δημοσίων συμβάσεων. Ε, ο ορισμός των κριτηρίων είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να βρει κανείς να ε, εντάξει αυτό το θέμα στη γενικότερη πολιτική. Τώρα, μια δεύτερη αρχή, και αυτό έχει να κάνει με τη συνθήκη, ε, είναι ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται και σε διοικητικό επίπεδο και τα πράγματα να μην ε, περιπλέκονται. Θα πρέπει κανείς προβληματιστεί κανείς σε, με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ανταγωνισμό. Ε, και οπωσδήποτε να καθοριστούν, καθοριστεί κάποιο κατόφλι. Συμφωνούμε για την απλοποίηση όσον αφορά τις επιχειρήσεις πρέπει φυσικά να δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπειρία. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και στην πράξη. Εγώ πιστεύω ένα ευρωπαϊκό θα λέγαμε διαβατήριο είναι πιο, πολύ χρήσιμο. Τώρα μια τελευταία παρατήρηση. Σαν ομάδα εμείς θα δούμε τι ακριβώς γίνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει ληφθεί μια απόφαση, αλλά θα πρέπει οι αποφάσεις οι δικές μας να θα πρέπει να υποβληθούν σε, μια ε, μελέτη ε, επιπτώσεων όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Να δούμε δηλαδή ποιο θα είναι το, ποια επίπτωση θα υπάρξει στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια οποιαδήποτε απόφασή μας. Υπάρχουν προσδοκίες από αυτό το χώρο. υπάρχουν κάποιες προθέσεις, κάτι το οποίο μπορεί να είναι καλό για τους μεν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι οριστικό σε αυτό το στάδιο. Να δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος της διαδικασίας και να δούμε ποιες θα είναι επιπτώσεις για τις μικροπιστές επιχειρήσεις. Πετυχαίνοντα μια απλοποίηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλβίνη. Ευχαριστώ κύριε θα ξεκινήσω από την τελευταία παρέμβαση. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι ε, οι δήμοι και οι κοινότητες, διότι πολλές φορές ε, μιλάμε για έναν δήμαρχο ο οποίος ε, ε, κάνει την ανάθεση, να δούμε, κατα... μάλλον είναι υπεύθυνο για, την, για τις αναθέσεις, για τις συνάψεις των συμβάσεων, ο δημόσιος ελεγκτής, άρα θα πρέπει και αυτούς να λαμβάνουμε υπόψη μας. Επίσης δεν είναι θέμα μόνο τιμής, δεν είναι χαμηλότερη προσφορά που θα πάρει την αγορά. Είναι θέμα, υπάρχει και το ποιοτικό κριτήριο, το κοινωνικό κριτήριο. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνο και τα υποστηρίζουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο στις ε, δημοτικές αρχές, στις περιφερειακέ αρχέ, για να δούμε πώ θα διαφυλάξουν με, τα, τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα των πολιτών και όχι μόνο να βλέπουν το οικονομικό όφελο. Επίσης, ε, η προσυπογραφή κάποιων δημόσιων, ε, ε, συγγνώμη, ε, διεθνών συμβάσεων, π.χ. του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, είναι σημαντικό. Επίσης ένα άλλο κριτήριο είναι η πρόθεση της τοπικής παραγωγής. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ε, πολιτική, όχι απλώς μόνο για να πλουστεύουμε τα πράγματα, άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι μια και ζούμε μια οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βοηθάει τους παραγωγούς που παράγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ελπίζω ότι θα ε, ε, γίνει αντιληπτό όχι μόνο σαν εμπόδιο ή σαν κόλλημα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Εμείς ε, πρέπει να κάνουμε και επιλογές, να μην είμαστε μόνο λογιστές. Επίσης τώρα η κατανομή σε ενότητες εργασιών, σε παρτίδες όπως είπαμε ε, είναι κάτι το θεμητό διότι εκτός από γιατί κάποιες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κάτω από κάποιο κατόφλι δεν μπορούν να συμμετέχουν άρα αυτή η κατανομή σε παρτίδες σε ενότητες εργασιών είναι κάτι το εφικτό δηλαδή επίσης χρειάζονται και υπεργολαβίες διότι ούτως ή άλλως θα χάσουμε τον έλεγχο Επίσης, επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάποια άλλα θέματα, να, οι οδηγίες ε, να εφαρμοστούν, ε, υπάρχουν ε, η, ας πούμε, η οδηγία για τις καθυστερούμενες πληρωμές. Η Ιταλία δεν την έχει, έχει εφαρμοστεί. Η Λομβαρδία ε, πληρώνει μέσα σε 90 μέρες η, το Ρέτζο Καλάμπρια χίλιες κάτι μέρες. Δηλαδή τώρα πώς θα εφαρμοστεί αυτό, αυτή η οδηγία στην Ιταλία δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ε, υποβάλαμε μια τροπολογία όπου το, λέμε ότι το κράτος θα πρέπει να εγγυώνται την φερεγγιότητα των ε, αρχών που πληρώνουν. Τώρα, στην, στην Καλαβρία δεν ξέρω από 1500 μέρες πώς θα περάσουν σε 90 ή σε 60 μέρες. Αυτό το θεωρώ λίγο ουτοπικό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ε, φερεγγιότητα και να είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζονται τα πράγματα τα οποία απαιτεί κάποια οδηγία, για πριν πω και η προηγούμενη οδηγία. Λοιπόν, τώρα, δεν θα ήθελα η ταχύτητα να ε, επιδεινώσει την κατάσταση και να ε, θίξει την ποιότητα των διατάξεων. Δηλαδή, μία-δύο εβδομάδες παραπάνω στη σκέψη δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους ε, δημάρχους μας ή στις αρχές που πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για και τον εισηγητή. Όντω έχετε δίκιο και για την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε. Οι συντονιστές, να το παρακολουθήσουμε κιόλας. Λοιπόν, οι συντονιστές σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουν το χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πετύχουμε την βέλτιστη ποιότητα στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να καλωσορίσω και μια ομάδα επισκεφτών που ήρθε από το Χάσιλτι, η κυρία Βάιλε της τους ε, κάλεσε. Πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τις ε, 10.30, διότι εκεί θα υπάρχει και μια ανταλλαγή απόψεων ε, για, με τους εμπειρογνώμονες. Λοιπόν, έχω 7 άτομα στον κατάλογο. Θα ήθελα να σας πω ποιοι είναι. Juvan, Mr. Schwab, Mrs. Styler, Mrs. Weiler, Mr. Meyer, Mrs. Schaldemoser. Can I just see if anyone else wants to join the list? Um... Κάποιοι άλλοι θέλουν να προσθεθούν. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να πάρει το λόγο. Λοιπόν, δύο λεπτά το περισσότερο. Ζητώ συγγνώμη που πρέπει να πιεστούμε και να, και να βιαστούμε, αλλά θέλω να δώσω και λίγο λόγο και στον εισηγητή και ο κύριο Βίνερ να θέλει να κάνει δύο σχόλια. Λοιπόν, δύο λεπτά ο καθένα. Ακούσαμε όλου του σκιώδεις ε, από, ε, από πλευράς των ομάδων. Λοιπόν, ασχολήσουμε την κυρία Κέπχαρτ. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, <coughs> Μεγάλε ευχαριστίες στο Μάκτα Ραμπέλα για την εξαιρετική πραγματικά δουλειά που κάνει και έκανε. Εδώ έχουμε ένα σημαντικότατο θέμα και ω συντονίστρια της σοσιαλδημοκρατική Ομάδας θα ήθελα αμέσω εδώ να πω ότι και εγώ θέλω η ποιότητα να είναι η μέγιστη προτεραιότητα και φυσικά για την ομάδα μα <coughs> θα πρέπει να αυτό να το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Και ο εισηγητής ε, και οι σκιώδεις εισηγητές αν χρειάζονται περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερη διορία δεν έχω καμιά αντίρρηση σε σχέση με την ε, ε, επέκταση. Θέλουμε να κάνουμε καλή δουλειά και αν χρειάζεται αυτός ο χρόνος είναι σαφές ότι πρέπει να εγκριθεί. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ομάδα μας γι' αυτό. Μια παρατήρηση εκ προημίου θα ήθελα να κάνω. Και εγώ θέλω να απλουστεύσουμε και εγώ θέλω να ανακουφίσουμε τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ποιότητας όμως. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε με ιδιαίτερο τρόπο το τι θα γίνει. Και όλα αυτά δεν σημαίνουν απορρίθμιση βέβαια, που στο τέλος τέλος μπορεί να αποβαίνει κατά της ποιότητας, εις βάρος της ποιότητας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση εκ προημίου λοιπόν και με το, με το πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο βέβαια, αλλά πρέπει να παρεμποδίσουμε οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις τρύπε ε, και τα παράθυρα που υπάρχουν νομοθετικά όσον αφορά τις συμβάσεις και να, τις... να παρακάμπτουν τις διαδικασίες και τους κανονισμούς. Γι' αυτό είναι σημαντικό το θέμα. πόσοι υπεργολάβοι θα εντάσσονται σε αυτές τις υποχρεώσεις. Και αυτό έχει τεράστια σημασία στο τέλος τέλος. Ώστε και εκεί πάλι τα κριτήρια από όλους να ισχύουν με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με τον καθορισμό των δημόσιων συμβάσεων. <clears throat> Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο για μένα. Φυσικά πρόκειται για την πιο ευνοϊκή προσφορά και φυσικά πρέπει να συζητήσουμε και τα κριτήρια τα οποία θα συναρτώνται με αυτή την πιο ευνοϊκή προσφορά να κινδύνου, να μην περιορίσουμε υπερβολικά το πλαίσιο εναντί αυτού που έχουμε σήμερα. Και ακριβώς η κοινωνική αηφορία, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική υπόθεση, θα πρέπει να μπορεί να διασφαλιστεί. Αυτά ήθελα και μπορώ να πω σε δύο λεπτά. Θα είχα και άλλα θέματα να καλύψω, αλλά ο χρόνος πιέζει και γι' αυτό εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Ah, thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κέφχαρτ. Α, έχασα τον κατάλογο μου. Ποιος είναι ο επόμενος. Ο κύριος Σβάμπ. Ο κύριος Σβάμπ, ευχαριστώ πρόεδρε. Και πάλι φυσικά από πλευράς μου ευχαριστήσεις για όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο με αυτόν τον πολύ εξαιρετικό τρόπο. Θα πρέπει οι συντονιστέ να αποφασίσουν το απόγευμα τι θα κάνουμε. Είναι παρόν το θέμα στην νομοθετική αυτή περίοδο και στη συζήτηση όλοι συμφώνησαν σήμερα να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να ενισχύσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά, να υπάρχει ελαστικότητα για όσου εμπλέκονται. Μα εκπλήσει ότι οι τροπολογίε σε λεπτομέρειε αντιφάσκουν μεταξύ του. Γι' αυτό έχει, σημαντική, έχει σπουδαιότητα το θέμα να δούμε ποιε είναι οι πλειοψηφίε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο στο τέλο να συνενέσουμε και να συμφωνήσουμε επί κάποιων προτάσεων. Όσα ακούσαμε δείχνουν ότι με όλη την κατανόηση που υπάρχει για τις δυσκολίες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και για τα θέματα τα κοινωνικά για τις δημόσιες αυτές συμβάσεις θα πρέπει στο τέλος τέλος να αναζητήσουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Το θέμα είναι διαδικαστικό. Θέλουμε το δυνατόν πιο γοργά, πιο γρήγορα να ολοκληρώσουμε ή θέλουμε γενικά να συζητήσουμε ε, για ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά θα πρέπει να δούμε ότι χρειάζονται ε, συγκεκριμένοι συμβιβασμοί και προτάσεις για να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα. Και από πλευρά του εισηγητή θα πρέπει να υπάρξουν και συμβιβαστικές προτάσεις επί των διαφορετικών αυτών πτυχών. Νομίζω σχετικά γοργά μπορούμε να καταλήξουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε λύσεις και θα χαιρόμουν αν το καταφέρναμε. Σε ένα σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στην κατηγορία 10, κλάστερ 10, για το θέμα της δημόσιας συνεργασίας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εδώ συνιστώσεις η κάθετη και η οριζόντια συνεργασία. Εγώ θα έλεγα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ομολογία που έχει ήδη θεσμοθετήσει να προσαρμοστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε λειτουργικοί. Και θα αναφερόμουν ρητά στην τροπολογία 63 και άλλες αλλά και στην ε, ε, αντίστοιχη τροπολογία που πρέπει να καταλήξουμε επ' αυτή σε συμβαστική τροπολογία όλοι. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα. Είναι δύσκολο το έργο του και καταλήγει σε ένα στάδιο το οποίο μας δίνει ένα τέτοιο, τέτοιο επίπεδο που δημιουργεί μια διαφάνεια Σίγουρα υπάρχει, έχουμε μια, ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Τώρα για τις τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να πω για το αναλογικό έλεγχο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός πολύ σαφής. Έχουμε να κάνουμε με τις ε, δημόσιες μεταφορές και τους ε, ταξιδιώτες. Υπάρχει το θέμα των, των δραστηριοτήτων των 90% Εγώ θα ήθελα να ακούω εδώ τι αφορά αυτό το ποσοστό. Τα γεύματα στις καντίνες έχει να κάνει με αυτά που είναι, ε, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι πολύ περίπλοκο. Μπορεί φυσικά να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε άλλες λεπτομέρειες. Το άρθρο 72 θα πρέπει να δούμε το, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές κοινότητες επίσης για τα θέματα που αφοράν την επιπτώσεις που θα έχει στο μέλλον στην αγορά θα, θα πρέπει να δράσουμε. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό με παράνομο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία στο μέλλον θα επανέλθω. Απλώς, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω με το εξής ε, ότι το κείμενο αυτό κα, καθ' αυτό ε, δεν θα έχουμε ένα κοινό κείμενο, θα είναι λάθος. Ε, θέλουμε να κάνουμε το, τα, οι δημόσιες προσφορές τώρα εδώ πέρα είναι ένα θέμα που έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι επιχείρηση. Δεύτερον, υπάρχουν πολλοί ορισμοί οι οποίοι θα πρέπει να είναι κοινοί. Δηλαδή σε ένα πρώτο κείμενο να έχουμε ένα α ορισμό και ένα β ορισμό λίγο αργότερα σε κάποιο άλλο σημείο δημιουργεί σύγχυση. Όταν μιλάμε για οριζόντια συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό ορισμό για να καλύψουμε τη νομική πτυχή. Θα πρέπει δηλαδή, είναι σίγουρο, να δουλέψουμε μαζί, από κοινού. Ευχαριστώ. Okay. Ξέρω ότι στενά συνεργάζεστε με τον κύριο Ταραμπέλα. Και επίσης ε, σε αυτό το πλαίσιο και για την δική σας έκθεση που εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται πρόοδος λοιπόν. Η κυρία Στάιλερ, μετά η κυρία Βάιλερ, μετά η κυρία Μάιερ και μετά Σάλτε Μόζερ. Η κυρία Στάιλερ παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ φυσικά και προς τον εισηγητή επίσης. Και στις 7 Σεπτεμβρίου είχαμε με πολύ επιτυχή ένα πολύ επιτυχέ σεμινάριο για τις ε, δημόσιε συμβάσεις και αγορές ε, στο Βούργο και ήταν ε, η πρόοδο πραγματικά εντυπωσιακή. ένα από του ομιλητέ ανέφερε και αυτό εντυπωσίασε σε σχέση με το έργο μας το ότι ο τρόπος με τον, αγοράζει, οποίο αγοράζει κανείς ε, καθορίζει πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε. Και για τις ε, τροπολογίες ε, που έχουν κατατεθεί υπάρχουν και τα κοινωνικά κριτήρια, το δίκαιο εμπόριο, η προστασία των εργαζομένων, η προστασία των διαφόρων αυτών εργαζομένων, η πρόθεση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα στα, στα πλαίσια της αποτελεσματικής αποτελεσματικότητα. Άλλοι αναφέρθηκαν στην απλούστευση και αποτελεσματικότητα. Ο χρόνο πιέζει. Διασυνδέονται όλα αυτά σε σχέση με τι παρατηρήσει εκείνων που δεν είναι αισιόδης εισηγητέ. Πολλοί από εμά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Κατέθεσα 13 τροπολογίε και θέλω να προχωρήσουν στι συζητήσει που θα διεξάγονται. Θα ήθελα να ζητήσω, Πρόεδρε, η διαδικασία για τα 10 αυτά κλάστερ, τι κατηγορίε αυτέ να τεθούν στο διαδίκτυο και να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα το Νοέμβριο. Ε, ίσως εδώ πρόκειται και για κάποια ε, χρονική, κάποιο χρονικό περιορισμό. Η και το επαρκέ πλαίσιο έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Περιορίζομαι σε αυτά στα δύο λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστώ και συμφωνώ πολύ μαζί σα. Και οι σκιώδεις συζητητέ συμφωνούν μαζί σα. Έχουμε ένα κοινό έγγραφο εργασία, ε, στο οποίο η ανάλυση των τροπολογιών θα πρέπει να γίνει και να διατεθεί αυτό σε όλα τα μέλη στο διαδίκτυο μετά συνεδρίαση ώστε να διευκολυνθούν. Όλοι και όλοι οι σκιώδεις ε, με ανοιχτό πνεύμα ε, προσεγγίζουν αυτέ τι διεργασίε όσον αφορά και τι δικές σα τροπολογίε. Η κυρία Βάιλερ επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ μόνο σε δύο θέματα, Πρόεδρε. Αλλά εκ προημίου θέλω να πω, δεν έχω πιστεί ακόμα δεν έχω πιστεί ακόμα ότι σε ένα τέτοιο τεράστιο, μια τέτοια τεράστια στίβα τροπολογιών μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό νομοθετικό έργο. Πολλή δουλειά θα απαιτηθεί από την ε, ε, νομική υπηρεσία και από τους συναδέλφους για να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν είναι υποχρεωτικά θετικό ότι η κοινοβουλευτική μας επιτροπή καταλήγει σε τόσες υπερβολικά πολλές τροπολογίες. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. 2.000 περίπου τροπολογίες. Υπερβολικό αριθμό. Δεν θεωρώ ότι εξυπηρετεί την υπόθεσή μας σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό ως εκ παρατήρηση. Δεύτερο τώρα. Συνάδελφε Ρούιλε, αγαπητοί συνάδελφε, πρέπει να προσέλθουμε και σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα στη δήλωσή σας και με τη διατύπωση ότι πρέπει να είμαστε λογικοί και να τηρούμε τις λογικές αναλογίες και συσχετισμούς και εγώ ε, προσεγγίζω θετικά αυτή τη φιλοσοφία αλλά πολλές φορές γίνονται υπερβολές ε, στην Γερμανία και αλλού αλλά δεν θέλω να αναφερθώ στη Ρουμανία και σε άλλα κράτη στα μεγάλα κράτη μέλη όπου γνωρίζουμε το τι γίνεται με το δικαίωμα συμβάσεων ήδη τώρα χρησιμοποιείται η δυνατότητα της πιο ευνοϊκής ε, οικονομικά προσφορά. ανεξάρτητα από το ότι μπορεί να υπάρχει συνένεση από όλους ότι δεν πρέπει πιο φτηνή προσφορά να υιοθετείται υποχρεωτικά. Πολλοί ξέρουν ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά λοιπόν με κάτι τέτοιο και αυτό δεν είναι τελικά η πιο ε, θετική προσφορά στο τέλος τέλος. Τώρα, αν κατάλαβα καλά από τη μετάφραση, εσείς κυρία Ρούλε θα θέλατε λέει να διαγραφεί αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια. από Αποκινούμε αυτό. Δεύτερον, υποτιμούμε τους εμπλεκόμενους στους στρατηγικούς στόχους. Εν τω μεταξύ η συζήτηση στο σύνολο της Ευρώπης, αλλά και πέρα από την Ευρώπη και σε άλλες υπήρους, είναι αυτονόητο ότι συμπεριλαμβάνει κοινωνική κριτήρια. Δεν είναι κάποια καινοτομία αυτή. Έχουν συνηθίσει αυτό το γεγονός πολλοί σε άλλα μέρη, στη Γερμανία υπάρχουν αυτά τα στοιχεία των κοινωνικών αυτών προδιαγραφών στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν είναι τίποτα καινοτόμο και καινούριο ο τα πολυάριθμα κριτήρια θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αν συμφωνήσουμε σε μία μη υποχρεωτική δέσμευση. Θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο και είναι ε, εφικτό νομικά να τα καταφέρουμε ώστε να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα στο τέλος τέλος. Έτσι, ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ κύριος Μάιερ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η οδηγία στρέφεται στα κράτη-μέλη για την υλοποίηση ουσιαστικά. Όμως οι τελικοί καταναλωτές, ε, δηλαδή ε, οι μικρομεσαίοι δήμοι κοινότητες τουλάχιστον στη δική μας περιφέρεια, και όταν έχουμε μεγάλες ε, τέτοιες για παράδειγμα ε, συμβάσεις όπως ε, το μεγάλο αεροδρόμιο του Βερολίνου οι περισσότερες όμως προσφορές αφορούν περιοχές με 5, 10, 20.000 το πολύ κατοίκους. Θέλουμε να στραφούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν και διαρωτώμενοι ποια είναι η επιβάρυνση στη σημερινή χρονική συγκυρία να συμμετέχει κανείς σε τέτοιου είδους προδιαγραφές ξεπερνά κατά πολύ τις δυνάμεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε συνήθισαν αυτή την επιβάρυνση και μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Πρέπει να υπάρχει μείωση επιβαρύνσεων και μείωση φόρτου ει βάρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδου προσφορέ για δημόσιε συμβάσει. Περί αυτού πρόκειται και γι' αυτό προτείνω να έχουμε μια συζήτηση επαϊόντων, ειδικών, όχι καθηγητές και νομομαθείς και τους παρόμοιους, αλλά κανονικούς πολίτε πολίτες, απλούς πολίτες που ζουν σε μεσαίες, πολίτες, σε μεσαίες πόλεις, με συγχωρείτε, μικρές και μεσαίες πόλεις και που εκεί πρέπει να γίνεται η προσπάθεια με 20, το πολύ 60 συνεργάτες να αντιμετωπίζουν αυτό το φόρτο εργασίας και να δουν και να μας πούν τι πρέπει να βελτιωθεί και τι μπορεί να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρία Σάντε Μόζε, παρακαλώ τώρα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους εισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές. Πραγματικά δεν σας ζηλεύω, πολύ δύσκολο το έργο σας. Πάντως ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει το ενδιαφέρον για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και αυτό πρέπει να μας ικανοποιεί γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και για μας και για τους πολίτες. Δεν σας ζηλεύω όμως, το επαναλαμβάνω. Να συμφωνήσω με την κυρία Στάιλερ για την διαδικασία εδώ στην Επιτροπή Καταναλωτών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, γιατί επιτρέπει και σε εμά που δεν είμαστε σκιώδεις να συμμετέχουμε. Γι' αυτό ε, σας ζητώ, απευθύνω μια έκκληση, να ξεκινήσετε με τις συμβαστικές τροπολογίες, να περιοριστεί ο αριθμός των τροπολογιών, για να δούμε σε ποιους τομείς μπορούμε να προχωρήσουμε, να συζητήσουμε, να επιτευχθεί η συμβαστική λύση ή θα, τι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ανοίξτε τη διαδικασία, ε, επιταχύνετε τα πράγματα, να καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά τι να σας πω Επίσης, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των κατοφλίων. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο αυτό το θέμα, διότι είχαμε με τους εμπορικούς μας εταίρους αυτή τη συμφωνία για τους κατόφλοι. Ίσως να είναι το θέμα δανέζικο, αλλά γιατί, γιατί δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα κατόφλια. Θα ήταν ένας εύκολος τρόπος για να είναι λιγότερη γραφειοκρατία για τις τοπικές αρχές. Επομένως, σας ρωτώ, σας ζητώ μάλλον για άλλη μια φορά να προσπαθήσετε να συζητήσετε αυτό το θέμα και μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όντως πρέπει να έχουμε ανοιχτό, ε, ανοιχτή διαδικασία, ανταγωνισμό, αλλά να ανοίξει η διαδικασία. Δεν σας ζηλεύω, επαναλαμβάνω και σας εύχομαι καλή τύχη. Ωραία, ευχαριστούμε όλους για την ε, συζήτηση και η κυρία Σάντερ, Σάντερ Μόζερ έχει απόλυτο δίκιο ότι θα πρέπει να ε, μοιραστούν οι συμβαστικές ε, τροπολογίες. Αυτό το συζητήθηκε και στους σκιώδεις συζητητές. Λοιπόν, η Κομισιόν, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να κάνετε μια μεγάλη παρέμβαση. Ε, ο κύριος Ταραντέλα θα είναι μετά. Ναι, ναι, ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση. Είναι η ίδια συζήτηση που έχουμε και στο Συμβούλιο. Ε, τα πράγματα ε, θα είναι πιο, πιο γρήγορα στο Συμβούλιο. Τέλος Οκτωβρίου, τέλ, αρχές Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκεί. Θα είμαστε έτοιμοι κι εσείς όποτε είσαστε για τον Τρίλογο. Αυτά. Ευχαριστώ. Για τα θέματα των κατοφλίων θα το συζητήσουμε ξανά, γιατί όντως είναι περίπλοκα διεθνή θέματα εδώ που θίγονται. Χαίρομαι που ο κατάλογος, ο, συγγνώμη, ο, τα έδρανα του Συμβουλίου είναι γεμάτα σήμερα. Σας καλωσορίζω. Κύριε Ταραμπέλα, σαν εισηγητής, μήπως θέλετε να μας, κάνετε τα, να μας δώσετε τα συμπεράσματά σας, επί του παρόντος τουλάχιστον. Ίσως να έκανα μια σύντομη παρέμβαση, Πρόεδρε, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε όσα ελέγχθησαν, ήταν πάρα πολλά. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της ομάδας μου, διότι έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ε, είναι στο χέρι, είναι ελεύθερος ο καθένας να το πράξει. Ε, έχουμε 1500 και τροπολογίες, δείχνει δηλαδή ότι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά πολύ κόσμο. Είναι λογικό να έχουμε 19% του ΑΕΠ σε Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αφορά αυτός ο τομέας και φυσικά πολλοί ενδιαφέρονται και καταθέτουν τροπολογίες. Και λέω ε, ευχαριστώ τις, τους της ομάδας μου είναι γιατί υπάρχει μια συνοχή στις τροπολογίες που έχουν καταθέσει. Έχω συνεργαστεί με τους ε, σκιώδεις συζητητές, ε, ε, εμείς υπε της ουσίας είμαστε και άλλες 7 επιτροπές ε, δραστηριοποιούνται για αυτή την οδηγία. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε διάφορα θέματα. Ε, θα μπορούσα εδώ να πω ότι ο ε, λοχαγός Σουάμπ έσωσε το στρατηγό Έγκελ. Το... Εγώ, ε, απ' τη μια μπορεί να είμαι κοντά στην κυρία Πέτικαν, και έχω και ένα συμπατριώτο μου και από αυτός κατέθεσε τροπολογίες τις οποίες συμμερίζουμε εν γέννη ε, είναι, όσο πιο ευρύ η ευρεία είναι μια ομάδα είναι τόσο πιο δύσκολο να ε, συντονίσει τι τις αυτά έχει η δημοκρατία όμως. Αλλά μην πάμε και σε αναρχία. Θα πρέπει δηλαδή να καταλήξουμε αργά ή γρήγορα σε συμβιβασμό. Φυσικά όλα δεν θα συμπεριληφθούν, δεν θα τα κρατήσουμε τις ορπολογίες. Θα πρέπει να περάσουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Ε, η κυρία Μπρίλιο, δεν ξέρω κάποιος άλλος, είπε ότι, ότι μας ζητάνε να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Απ' την άλλη πρέπει να αποφύγουμε το, το θέμα της παγίδας της χαμηλότερης τιμής. Ε, ε, υπάρχουν νέες αντιλήψεις, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διατηρήσουμε το στόχο μας ή μη οδηγούμαστε σε περιπέτειες σε περίπλοκες καταστάσεις. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Τώρα, για το θέμα της κοινωνικής βιώσιμης διαδικασίας, τι ακριβώς είναι. Φτιάξτε. Είναι μια αρχή η οποία θέλει να σεβαστεί κάποιους κανόνες διεθνείς, ε, συμβάσεων σε, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο για το θέμα της εργασίας. Συμβάσεις συλλογικέ που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά δικαιώματα, συνθήκες εργασίας και αυτή η αρχή φυσικά θα πρέπει ίσως να εφαρμοστεί και στα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των δημοσίων συμβάσεων. Κριτήρια ε, με τα οποία αποκλεί κανείς ή δέχεται κανείς κάτι. Ε, έχουν να κάνουν εδώ πέρα με ένα ε, ψηφιδωτό. Και συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε. Από τη, μια, τη μια προσπαθούμε να είμαστε πολύ ακριβοί, ακριβόλογοι σε θέματα ε, και αυτό ίσως να οδηγεί σε γραφειοκρατία, αλλά ε, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. ανέφερε κάτι ο Σαρδίνη. Μας οδηγεί σε χροκοπία με τα στοιχεία που μας έδωσε. Φερρυπίν, υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε βάζουμε μια προθεσμία να πληρωθ... γίνουν οι πληρωμέ μέσα σε 30 μέρε, Φερρυπίν. Ε, θα κλείσω τώρα, κύριε Πρόεδρε. Απ' τη μια, κανόνε που θα πρέπει ε, ε, γίνονται σεβαστοί, άλλου κάτι του οποίου θα αποφύγουμε. Φυσικά υπάρχει και αγγλοσαξονική προσέγγιση χωρί κανόνε. Εμεί τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, Να έχουμε κανόνε από τη μια, απλοποιημένοι από την άλλη και να έχουμε φυσικά και κυρώσει όταν χρειάζεται. Έχουμε την οικονομία, ξέρουμε ότι κάποιο δικαιούται να έχει μια σωστή εργασία, σε σωστή τιμή ένα προϊόν. Φυσικά, απ' την άλλη, πρέπει να γίνονται σεβαστοί, ε, σεβαστές συνθήκες εργασίας και οι σωστέ διαδικασίες. Να ευχαριστήσω τη, τη βεθό μου αριστερά και επίσης και το δεξί μου χέρι την κυρία Μπερτουλέση, η οποία είναι πολύ δραστηριοποιημένη στους ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Ε, να ευχαριστήσω επίσης ε, τους σκιώδες και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα σαφέστατο μήνυμα. Επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Με υποστήριξε μέχρι τώρα. Είχαμε και μια βίντεο διάσκεψη όταν είμαστε στο Στρασβούργο προσεγγίσαμε μια σειρά θεμάτων. Συμμετείχαμε όλοι και εύχομαι φυσικά να καταλήξουμε στα πλαίσια των προθεσμιών. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε γρήγορα. Συμμερίζονται αυτή την προσέγγιση και οι συνάδελφοι και η Επιτροπή. Και τώρα θα έλεγα αρχίζει η σύνθεση του έργου, του επίπονου έργου που έχω μπροστά Λοιπόν, πολύ καλά. σα ευχαριστούμε πολύ Μακταραμπέλα για τι κατευθύνσει που δώσατε για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ήταν μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σήμερα το πρωί. Θα περάσουμε στην εξέταση των λεπτομεριών πιο εξειδικευμένα με πολύ προσεκτικό τρόπο. Ευχαριστώ. Όσοι δεν παραμείνουν για την επόμενη υπόθεση ανταλλαγή απόψεων με του επαΐοντες να εγκαταλείψουν την αίθουσα ήσυχα, διότι θέλω να προχωρήσουμε στη συνέχεια και αν θέλει κάποιο να συμπεριληφθεί επίσης στην ανταλλαγή απόψεων. Εντάξει, λοιπόν. Le... Λοιπόν, παρακαλώ, ζητώ από όλους όσους δεν θέλουν να παραμείνουν για αυτή την ανταλλαγή απόψεων στο επόμενο σημείο να μας αφήσουν να συνεχίσουμε. Κάποιοι εκεί πίσω θέλουν να βρουν μια θέση να καθίσουν. Καθίστε, αν βρείτε θέση, αυτό θα είναι καλό. Παρακαλώ. Good. Πολύ καλά, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζω λοιπόν στο δεύτερο αντικείμενο ως θέμα της σημερινής μας πρωινής συνεδρίασης. Συζήτηση με τους επαΐοντες για την απόσπαση εργαζομένων, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διασυνοριακή συνεργασία και η συμμόρφωση. Συντάσσουμε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης ε, εμείς και έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα αυτό για μας στο πλαίσιο της του έργου για την ενιαία εσωτερική αγορά και για την λειτουργία, λειτουργικότητα της ενιαίας εσωτερική αγοράς. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια κυρία Τούρουνεν, διότι έχει μπορέσει να ε, συνενώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα επαϊόντων. Προσβλέπουμε στο να ακούσουμε τις απόψεις σας σήμερα το πρωί. Στους φακέλους σας πρέπει να έχετε ένα αντίγραφο του προγράμματος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα πλήρη βιογραφικά και τα στοιχεία για τους επαΐοντες. Δεν θα σας τα διαβάσω αυτά σε λεπτομέρειε. Τους καλωσορίζω καθώς θα λάβουν τον λόγο να μας προσφωνήσουν. Είναι ευπρόσδεκτοι. Ξεκινώντας για την ε, έναρξη αυτής της συνάντησης επαϊόντων και για να θέσουμε εδώ το πλαίσιο αυτών των θεμάτων. Θα λάβει τον λόγο η κυρία Τούρουνεν. Εισαγωγικά θα κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Μετά οι επαΐοντες θα έχουν 10 λεπτά ο καθένας. Και μετά θα έχουμε τον λόγο που θα δοθεί στους γενικούς εισηγητές ε, και όλοι να σχολιάσουν τα όσα θα έχουν ακούσει και στο τέλος θα σχολιάσει η κυρία Τούρουνεν ολοκληρώνοντας. Σας δίνω τον λόγο εισαγωγικά λοιπόν κυρία Τούρουνεν για να έχουμε την έναρξη αυτής της ακρόασης επαϊόντων. Η κυρία Τούρουνεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που προσήλθατε σήμερα σε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα κάποιες γενικές παρατηρήσεις να κάνω σε σχέση με αυτή την πρόταση. Τι έχουμε μπροστά μας ως πρόταση κάπως. Τι αναμένουμε από τους επαΐοντες ε, πώς θα μπορούν να μας διαφωτίσουν και να μας ενημερώσουν και στο τέλος κάποιες εισαγωγικές σκέψεις και παρατηρήσεις για το τι θα γίνει την Παρασκευή, όπου έχουμε την τελική προθεσμία για την έκθεσή μου από το χρονοδιάγραμμα. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι φυσικά ακρογωνιαίος λίθος της Ευ... Ευρωπαϊκής Ενιαίας Εσωτικής Δίνει το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες να μετακινούνται ελεύθερα και να υπόκεινται σε ίση μεταχείριση σε σχέση με άλλους εργαζόμενους σε σχέση με το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, με του εργαζόμενου ενό συγκεκριμένου κράτου μέλου. Επίση, η ελευθερία παροχή υπηρεσιών είναι θεμελιώδη ακρογωνίω λήθο για την εσωτερική αγορά. Δίνει το δικαίωμα σε επιχειρήσει να παρέχουν υπηρεσίε σε κράτη-μέλη. Οι επιχειρήσει μπορούν επίση να αποσπούν του εργαζομένου του σε ένα τέτοιο κράτο μέλο. Και αυτό θα αφορά τη σημερινή μα συζήτηση σήμερα και τους επόμενους ε, μήνες προσεχώς. Για να ρυθμιστούν όλα αυτά για την, έχουμε την οδηγία της απόσπασης εργαζομένων 96-71. Ωστόσο όμως, παρακαλώ λίγη ησυχία. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Γίνεται αυτό. Μας ενοχλεί η φασαρία και οι συνομιλίες σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έλεγα, αυτή η οδηγία ήταν ανεπαρκής όπως καταδείχθηκε. Ιδιαίτερα έχουμε νομολογία από πλευράς του, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που οδήγησε σε συζήτηση η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των θεμάτων αυτής της οδηγίας και του ρόλου των συνδικάτων για το, τα δικαιώματα των αποσπόμενων εργαζομένων. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα, σε αυτό το πλαίσιο. Διότι σε κάποια κρατημέλη ζούμε, βιώνουμε προβλήματα με την απόσπαση και οι κανόνες για την απόσπαση, οι κανονισμοί δεν γίνονται σεβαστοί. Υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σχέση με εργαζόμενους ενός κράτους μέλους και εργαζόμενους από άλλα κράτη-μέλη που προσέρχονται σε αυτό το κράτος να εργαστούν. Βλέπουμε παράκαμψη και αποφυγή συμμόρφωσης και βλέπουμε προβλήματα όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύτατο φάσμα προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για μια οδηγία συμμόρφωσης το Μάρτιο. Η ιδέα είναι να θεμελιώσουμε στην υφιστάμενη οδηγία και να διασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί στην οδηγία 96-71, οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται και θα είναι σεβαστοί. Και έτσι, αναφέρω παράθεμα, στοχεύουν όλα αυτά για να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της οδηγίας 96-71. Επίσης υπάρχει επιθυμία να θεσπιστεί ένα γενικό κοινό πλαίσιο για τα σωστά μέτρα και πιο κατάλληλα μέτρα για μια πιο ενιαία εφαρμογή και πιο αποτελεσματική εφαρμογή και συμμόρφωση με την οδηγία. Μέτρα επίσης για την αποφυγή οποιασδήποτε παράκαμψης ή κατάχρησης των κανόνων και κανονισμών. Σήμερα σας προσκαλέσαμε εσά για να μας προσφέρετε κάποιες σκέψεις σας για αυτή την πρόταση και επίσης για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή τι βλέπετε και βιώνετε εσείς ότι είναι προσκόμματα και εμπόδια στην καθημερινή σας δουλειά σε σχέση με αυτά τα θέματα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να κατανοήσουμε εμείς ε, αυτά τα θέματα. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα είναι γνωμοδοτούσα Επιτροπή. Υπάρχει ε, αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για αυτό το θέμα, όμως είναι σαφές για μας ότι αυτό το θέμα αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά. Γι' αυτό δίνουμε τέτοια σπουδαιότητα στα θέματα αυτής της οδηγίας εδώ στην Επιτροπή ΙΜΚΟ από πλευράς μας στη γνωμοδότηση. Τρία κυρία ερωτήματα που απευθύνονται σε εσά. Δηλαδή, υπό το πρίσμα της δικής σας ξεχωριστής δουλειάς, από την, τις επιχειρήσεις που προέρχεστε κάποιοι, από τις εθνικές αρχές που προέρχεστε κάποιοι άλλοι. Α, α, ποια εμπόδια και προσκόμματα, ποιες προκλήσεις βλέπετε πρέπει να αντιμετωπιστούν όταν έχουμε θέματα απόσπασης εργαζομένων. Τι χρειάζεται ώστε διασυνοριακά η συμμόρφωση και η επιβολή να είναι πιο αποτελεσματική και να γίνονται επιθεωρήσεις και ε, να υπάρχει εποπτεία ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που αναμένουμε να θίξετε και κάποιες πρώτες ιδέες από πλευράς μου ως κατευθυντήριες γραμμές για να ξέρετε πού στοχεύουμε εμείς με αυτές τις ε, δράσεις μας. Πρώτον, καλωσορίζουμε εμείς αυτή την πρόταση. Είναι σαφές ότι χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με αυτή την οδηγία. Δεν είμαι βεβαία βέβαια αν αυτή η οδηγία και η επιβολή της θα επιλύσει όλα τα προβλήματα και τις προσφυγές στα δικαστήρια και τις τριβές, προστριβές που υπάρχουν. Αν τα καταφέρουμε όμως, αυτά είναι μέσα και εργαλεία για να βελτιωθούν οι καθημερινές προϋποθέσεις συμμόρφωσης και εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Πρέπει να επικεντρωθούμε πρώτον στο να μεταθέσουμε το, το επίκεντρο προσοχής μας όχι μόνο στην ελευθερία και στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, δεδομένων αλλά και στην προστασία δικαιωμάτων τους. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τους περιορισμούς στα κράτη-μέλη για τα, ε, τις δυνατότητες εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με κάποια θέματα. Τουλάχιστον πρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό και όχι περιορισμένο κατάλογο. Μόνο έτσι θα είναι δυνατόν το δικαστήριο να λάβει υπόψη όλα τα θέματα τα οποία ε, ενέχονται εδώ. Δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε αυτό τον ε, κατάλογο και να παγώσουμε τις νομιμότητες οικονομικές εξελίξεις όσον αφορά τα πλαίσια επιβολής και συμμόρφωσης. Τρίτον, πρέπει να δούμε διάφορα πρότυπα από την αγορά εργασία. Στη Σκανδιναβία, στι σκανδιναβικέ χώρε, έχουμε ένα ξεχωριστό σύστημα. Έχουμε όμως σημαντικέ διαφορέ από κράτο σε κράτο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα διαφορετικά αυτά τα συστήματα θα είναι μεν σεβαστά, αλλά ταυτόχρονα τα συνδικάτα θα παίζουν ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο όταν ε, έρχεται η στιγμή να καθορίζουν τους όρους ε, συμμόρφωσης και σεβασμού, για παράδειγμα, συλλογικών συμβάσεων, αν δούμε τι γίνεται με άλλες χώρες. Τέταρτο, η συνεργασία των κρατών μελών πρέπει να είναι υποχρεωτική, γοργή και αποτελεσματική σε σχέση με τα πλαίσια αυτά. Πέμπτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ισοδίκαιο πλαίσιο για τον ανταγωνισμό. Να μην υπάρχει αν, ε, παράνομος, αθέμητος ανταγωνισμός όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες ε, ενδιαφέρουσες προοπτικές εδώ. Το άρθρο 12 για παράδειγμα ε, για τις, ε, τον κοινό επιμερισμό ευθυνών είναι ένα νέο σχετικά εργαλείο. Φυσικά θα πρέπει να είναι σεβαστές οι εθνικές διατάξεις μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Τελευταία παρατήρηση. Όλα αυτά, αυτή είναι μια οδηγία που ε, δίνει εργαλεία και μέσα για να αντιμετωπίσουμε την εξαπάτηση και τις ε, σκιώδεις ε, εταιρείε και άνομες και παράνομες πρακτικές. Αυτά όσον αφορά ιδιαίτερα και τους ορισμούς και το άρθρο 3 για την ε, αντιμετώπιση της παράκαμψης και αποφυγής συμμόρφωσης. Αυτές είναι κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Έχει μετατεθεί η ισορροπία των πραγμάτων μετά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έτσι πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή την ισορροπία ώστε να υπάρχει ένα ισοδίκαιο πλαίσιο ε, διαμόρφωσης πραγμάτων και δραστηριοποίησης για την ενιαία εσωτερική αγορά για την απόσπαση εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ακούσουμε τώρα τους εμπειρογνώμονές μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε άτομα εδώ παρόντα τα οποία ε, εμπλέκονται άμεσα στα θέματα αυτά, ε, αφορούν την, ε, το σεβασμό εργατικών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την επιθεώρηση εργασίας. Έχετε 10 λεπτά στην διάθεσή σας. Κάποιοι έχετε και διαφάνειες. Ε, Έχουμε, έχετε μοιράσει κιόλα ε, την, ε, την παρουσίασή σας, είναι διαθέσιμη η παρουσία σας. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Παύλο Πάραμο, ο οποίος εργάζεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και ασχολείται με την επιθεώρηση, τομέα επιθεώρηση εργασίας μετά θα ακούσουμε τον κύριο Φίλιπ Φον Τρόισεν, ο οποίος εργάζεται στην Γενική Διεύθυνση Τελωνίων, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Οικονομικών. Το Τελωνίο αναφέρε, ε, ασχολείται με θέματα δήλωτης εργασίας και εδώ θα μας μιλήσει για τον δικό του ρόλο. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Τόμας Μάγερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου των Πολωνών ε, εργοδοτών, θα ασχοληθεί με το θέμα από την σκοπιά των εργοδοτών και κατακλείδη ο κύριος Κλάς Μίκελ Γιόνσον, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των νομικών συμβούλων των, ε, της Συνομοσπονδίας ε, Σουηδικών Συνδικάτων. Θα μας μιλήσετε και για την δική σας εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Έμιλη που συγκέντρωσε όλο αυτόν τον κόσμο εδώ. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Πάραμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ και την εκπρόσωπο, την κυρία Τούρουνεν και τα, τους άλλους ευρωβουλευτές, μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τους βοηθούς. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να εκφράσουμε κάποιες απόψεις μας σε σχέση με το πρόβλημα της απόσπασης, προσωρινής απόσπασης εργαζομένων και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω το ότι η απόσπαση εργαζομένων είναι μια τάση ασταμάτητη που δεν μπορεί να σταματήσει στην Ευρώπη. Κάθε μέρα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων που αποσπώνται και μετακινούνται από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη προσωρινά σε άλλα. Και αυτό έχει σπουδαιότητα, είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι πρέπει να ληφθούν μια ολόκληρη σειρά μέτρων ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εθνικές νομοθεσίες να εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε ένα ενιαίο πλαίσιο σε αποτελεσματικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ο νόμιμο ανταγωνισμό και οι αρχέ του νόμιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Γιατί είναι ανάγκη να πάμε πέρα από τα πλαίσια τη οδηγία αυτή 96-71. Λοιπόν, πρώτον, επειδή οι διμερεί συμφωνίε δεν επαρκούν αφ' αυτών εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας μια και τα θέματα <clears throat> συνεργασίας δεν μπορούν να ρυθμίζονται από τα κράτη-μέλη αφ' αυτών αποκλειστικά και μόνο. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι η νέα νομοθεσία που εγκρίνεται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επίση είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ότι η έλλειψη, η απουσία συνεργασίας και η απουσία εφαρμογής του νόμου μπορεί να δίνει αφορμή σε περιπτώσεις απάτης, σε διάφορες περιπτώσεις και παραβιάσεων κανόνων. Ποιε είναι οι κυριότερε προκλήσει λοιπόν αυτή τη νέα νομοθεσία, χωρί καμιά αμφιβολία, είναι το να πετύχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ προστασία των εργαζομένων και τη ελευθερία παροχή υπηρεσιών. Να πετύχουμε μια πάγια, σωστή λειτουργία. Μια καλή λειτουργία του συστήματος ΙΜΗ, δηλαδή πληροφόρησης και συνεργασία και καλύτερη εφαρμογή όσον αφορά τι αρχέ τη οδηγία 96 96-71, καθώς και μια καλύτερη αμοιβαία συνεργασία και αρρωγή και δυνατή, δυνατόν να επιτευχθεί η αναγνώριση των κυρώσεων που θα πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων και παραβάσεων. Ε, μία από τι κύριε ε, τριβέ μπορεί να είναι το πώς θα καθορίζουμε τέτοιες άνομες, παράνομες περιπτώσεις όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων. Έχουμε δύο εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάζονται. Η θέσπιση κάποιων περιγραφικών στοιχείων για μια παράνομη τέτοια κατάσταση με ένα κλειστό πίνακα, με ένα κλειστό κατάλογο. Κάτι τέτοιο δημιουργεί ίσως μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα. Όμως ωστόσο τα δικαστήρια θα έχουν τα χέρια τους δεμένα όταν θα έρθει η ώρα να ερμηνεύσουν όλα αυτά και να καταπολεμήσουν τις παράνομες τέτοιες ε, έκδηλα παράνομες καταστάσεις. Η άλλη δυνατότητα είναι ένας ανοιχτός κατάλογος. Δίνει μεγαλύτερη ελαστικότητα. Τα δικαστήρια θα έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για την ερμηνεία τους και αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για την καταπολέμηση απατών. Ένα μείζον θέμα είναι τι θα γίνει όταν διαπιστώνεται μια παράνομη τέτοια κατάσταση κατάσταση στην απόσπαση ε, εργαζομένων. Θα εφαρμόζεται η οδηγία μόνο σκληρό πυρήνα συστάσεων. Θα εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτου προέλευση. Θα ε, εφαρμόζεται ο κανονισμό ε, Ρώμα 1 που θα είναι ω η υλοποίηση των συμβάσεων εργασία και ο σεβασμό του. Υπάρχουν πολλέ συζητήσει για αυτό το θέμα. Τρία θέματα είναι όμω βέβαια. Πρώτον, ότι η νομοθεσία κοινωνική ασφάλεια όσον αφορά παράνομε καταστάσει θα είναι εκείνη του κράτου προέλευσης. Αυτό καθορίζουν οι ξεχωριστοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση. Οι αποσπόμενοι εργαζόμενοι σε μια τέτοια περίπτωση απάτης δεν μπορούν να βρίσκονται κάτω από χειρότερες καταστάσεις απασχόλησης σε σχέση με τους εργαζόμενους που αποσπώνται μέσα στο πλαίσιο μιας νόμιμης τέτοιας απόσπασης. Ο αποσπόμενος προσωρινά εργαζόμενος με ε, τρόπο σε περίπτωση απάτης θα πρέπει να μπορεί να καθορίζεται όπως και ο ε, εργαζόμενος εκείνος σε περίπτωση παραβίασης όσον αφορά τον ε, κανονισμό αυτό της ε, Ρώμα 1. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες και η δυνατότητα να χρησιμοποιείται το ίμι. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν πέρα από τις αρχές μπορεί να εξεταστεί για εκείνες τις χώρες που ο έλεγχος ε, των συνθήκων εργασίας γίνεται από τους κοινωνικούς εταίρους σημαντικό θέμα και ενδιαφέρον θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να εντάξουμε αυτή την εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων μέσω του ΙΜΗ αν μπορούν να γίνουν μέσω μιας αρχής ή άμεσα μια αρχή εκπροσώπηση ή άμεσα ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Η ανταλλαγή απόψεων γίνεται μέσω του συστήματος ΙΜΗ. Επαρκεί αυτό ή πρέπει επίσης ε, να θεωρούμε ότι χρειάζεται οι αρχέ του κράτου να έχουν πρόσβαση σε μητρώα άλλων κρατών. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τι είδου μητρώα. Μητρώα εμπορικά ή μητρώα διοικητικά. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα προστασία προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που μπορούν να επιβληθούν, σε έναν πάροχο υπηρεσιών από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, πάλι τίθεται το εξή θέμα τριβών. Ανοιχτός κατάλογος ή κλειστός κατάλογος. Ανοιχτός κατάλογος υποχρεώσεων ή κλειστός ε, περιορισμένος τέτοιος κατάλογος υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει με αυτά που αναφέραμε προηγούμενα. Νομική βεβαιότητα ή μη νομική βεβαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης απάτης. Και κυρίως ε, πάνω απ' όλα, πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε εκείνα τα κράτη που έχουν συγκεκριμένα συστήματα ζητήματα συνδικαλιστικά. Για παράδειγμα, όπου η εργασιακή νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω εκπροσώπησης συνδικάτων για τις συλλογικέ συμβάσεις ε, με μεγαλύτερο ή μικρότερο εύρος ε, ρυθμίσεων για τις ε, συμβάσεις εργασίας. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πιθανή υποχρέωση να καθορίζεται ένα αρμόδιο άτομο για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι απαραίτητο αυτό. Μήπως είναι υπερβολική επιβάρηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις όχι. επίση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αναζητηθεί η σωστή ισορροπία για την αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των προβλημάτων. Όσον αφορά αυτές τις υποχρεώσεις πάλι, επίσης υπάρχουν κάποια συμπεράσματα. Ισότητα. Η ισότητα όρων όσον αφορά τις ε, κρατικές αρχές. Είναι ένα σαφές συμπέρασμα αυτό. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία είναι σημαντικά, όπως είναι τα έγγραφα τα οποία αφορούν και την ίδια την υγεία των εργαζομένων πολλές φορές και είναι σημαντικό μέσα στις απαιτήσει για τον πάροχο υπηρεσιών να μπορούν συμπεριλαμβάνονται αυτές οι διατάξεις αυτών των εγγράφων και για την κοινωνική ασφάλιση εξίσου. Και όταν κάνουμε λόγο για την, τον κλειστό κατάλογο ή ανοιχτό κατάλογο υπάρχουν εναλλακτικέ πιθανές τρίτες λύσεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ε, ομάδα του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά που μπορεί να θεσπιστεί μια ξεχωριστή διαδικασία ώστε να εγκρίνεται ένας ανοιχτός κατάλογος, από την άλλη πλευρά όμως να μπορούμε να κλείνουμε σταδιακά ένα τέτοιο κατάλογο ώστε να υπάρχει ένα, μια μεγαλύτερη ε, ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνεται για την προστασία των εργαζομένων. Όσον αφορά τα συμβατικά θέματα για επιχειρήσεις που είναι υπεργολάβοι Πάλι εδώ υπάρχει υποχρέωση αλληλεγγύης όσον αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις. Πράγματι, η υποχρέωση αλληλεγγύης όσον αφορά την υπεργολαβία είναι αποτελεσματική διάταξη, διότι μπορεί να είναι αποτρεπτική η διάταξη αυτή. Το συμπέρασμα είναι, το, συμπέρασμα θα, είναι, το, η επίπτωση θα είναι μεγαλύτερη σε κάποιες χώρες σε σχέση με άλλες, αν χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα επιπρόσθετα ένα άλλο θέμα που είναι και αυτό σημαντικό η εκτέλεση και η επιβολή διασυνοριακά των κυρώσεων. Τι γίνεται όταν παραβιάζει κάποια διάταξη μια επιχείρηση σε σχέση με το κράτος υποδοχής. Θα υπάρχει η κύρωση από πλευρά των αρχών αυτού του κράτους εις βάρος αυτής της επιχείρησης ή όχι. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει τίποτα. Μέχρι πρόσφατα είχε δημοσιευθεί μια μελέτη που είναι της ε, Επιτροπής Αρμοδίων της Επιθεώρησης Εργασίας που αποκλήθηκε θυμπέλες ε, υπό την ηγεσία της Ισπανίας αλλά υπάρχει και η συμμετοχή Γερμανίας, Ουγγαρίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Αυστρίας, Μάλτας, Ιταλίας. Τα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχει απόλυτη έλλειψη, απόλυτη απουσία εκτέλεσης και εφαρμογή των κυρώσεων. Δεν υπάρχει αναγνώριση των ε, ποινών και προστήμων και υπάρχει ο κίνδυνος ατιμορρησίας επιχειρήσεων στο τέλος τέλος. Και τέλος, τελευταίο, ένα άλλο σημαντικό θέμα και αυτό αν θα υλοποιείται η αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων μέσω του ΙΜΗ και την θέσπιση ενός εξειδικευμένου συστήματος διότι δεν είναι επαρκείς όλες οι αρχές, δεν βρίσκονται όλες στο ίμι και επιπλέον απαιτούνται διεργασίες, έντυπα, έγγραφα και η εποπτεία και η επιθεώρηση εργασιακή. Ευχαριστώ. thank you very much Mr. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πάραμο για, καταρχάς γιατί σεβαστήκατε το χρόνο, αλλά και γιατί μας δώσατε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις ε, και για τα θέματα που απασχολούν την κυρία Τουρούνεν. Λοιπόν, περνάμε τώρα στον κύριο Φον Πρόσιον και αυτός έχει 10 στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ για την ε, προσφορά και δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα πράγματα υπό το πρίσμα της Γερμανίας. Η Γερμανία είναι μία από τις μεγαλύτερες τρεις χώρες υποδοχής για τους εργαζόμενους, αποσπόμενους εργαζόμενους. Έχουμε πάνω από 15 χρόνια πείρας με την εφαρμογή του ε, πλαισίου απόσπασης εργαζομένων. Θα ήθελα σύντομα να φωτίσω λίγο το παρασκήνιο που οδήγησε σε αυτή την πρόταση που δεσμεύει τα κράτη-μέλη να δημιουργούν ελάχιστες προϋποθέσεις ε, που θα ισχύουν για τους αποσπόμενους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα <clears throat> ο εργοδότης θα έχει την έδρα του. Ελάχιστοι όροι απασχόλησης. Επίσης ε, και ελάχιστοι κανόνες για τον ελάχιστο μισθό, αναγκαίοι κανόνες. Η ίδια η οδηγία για την απόσπαση δεν έχει κάποιες προδιαγραφές για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, ε, αυτό το πλαίσιο προσεγγίζει αυτή η οδηγία. Δημιουργεί προδιαγραφές και όρους συνεργασίας μεταξύ αυτών των αρχών. Ποια είναι τα κυριότερα σημεία υπό το πρίσμα μας για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα διασφαλίζουν τους ε, όρους ελάχιστου μισθού και απασχόλησης που πρέπει να είναι σεβαστοί. Τα βιώματά μα από πλευρά πείρα πρέπει να υλοποιούν δύο κανονισμού. Πρώτον, στόχο πρέπει να είναι η συνεργασία για την υλοποίηση των ελάχιστων όρων απασχόληση που μπορεί να είναι ε, επιτυχής ο στόχος αν γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις στον τόπο εκείνο όπου παρέχεται η εργασία από τους αποσπόμενους εργαζόμενους είναι υποχρεωτική μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των στόχων και καθηκόντων του κράτους αποστολής και του κράτους υποδοχής. Για μας ε, υπό το άρθρο 7 του, της σημερινής διατύπωσης ε, δεν ε, επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Υπάρχουν εδώ κάποια κενά. Εδώ πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος θα διασφαλίζει την υλοποίηση των ελάχιστων όρων απασχόλησης και αυτό είναι στόχος των αρχών του κράτους υποδοχής που πρέπει να μπορούν να δραστηριοποιηθούν αυτές οι αρχές ανεξάρτητα και αυτοτελώς διότι το κυριότερο είναι οι όροι και οι ε, έλεγχοι στο κράτος υποδοχής. Μόνο τότε έχουν νόημα τέτοιοι έλεγχοι. Μόνο εδώ στο κράτος υποδοχής μπορούν να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι και να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις ε, ε, διασφαλίζουν ή όχι τους όρους αυτούς. Αυτό σύμφωνα με τα βιώματά μας εμπειρικά. Ε, ο στόχος έχει και πολύ ε, φιλόδοξους ε, όρους προϋποθέσεων και προθεσμιών για αυτή τη συνεργασία. Έχουμε και το θέμα της πρόσθετης εργασίας. Το άρθρο 3 στοχεύει στην αποφυγή παράκαμψης και μη συμμόρφωσης. Υπάρχουν εδώ και εξειδικευμένα τέτοια κριτήρια για την διασφάλιση απόσπασης. Ιδιαίτερα θα πρέπει οι εμπλεκόμενες στην αγορά επιχειρήσεις να διαφοροποιούνται από τις επιχειρήσεις που είναι σκιώδεις και διαθέτουν μόνο ένα ταχυδρομικό κυβότιο, μια ταχυδρομική θηρίδα μόνο ως διεύθυνση. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει αντιστοιχεία σε σχέση με τους όρους επιβολής. Αυτό είναι που απαιτείται, γιατί διαφορετικά η συνεργασία των ε, κρατικών αρχών δεν μπορεί να διασφαλίζει τους στόχους αυτής της απόσπασης. Θα μπορούσε σε αντίθετη περίπτωση να μην διασφαλίζει επαρκώς την προστασία των εργαζομένων. Και έτσι ο στόχος της ίδιας της απόσπασης και η προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται θα βρισκόντουσαν σε αντίφαση. Υπάρχει και ο κίνδυνος το άρθρο 3 να δημιουργεί μια επιβαρημένη δαπανηρή γραφειοκρατική διεργασία που δεν θα είχε καμιά πρόσθετη αξία για τους αποσπόμενου εργαζόμενους. Το σύστημα ΙΜΗ πληροφόρησης και ενημέρωσης που ακριβώς για το πεδίο εφαρμογής δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και μέσο συνεργασίας. Το ΙΜΗ όμως δεν μπορεί να έχει αποκλειστικό χαρακτήρα και περιοριστικό χαρακτήρα και άλλες μορφές και τύποι διακρατικής συνεργασίας πρέπει να, μπορεί να, να μπορούν να διασφαλίζονται. Αυτό ιδιαίτερα και για διμερείς συμφωνίες Πρέπει να είναι δυνατόν μεταξύ ήμι και άλλων μορφών συνεργασίας να υπάρχει εναλλακτική χρήση και επιλογή. Δεν υπάρχουν παντού τα ίδια προβλήματα και ίδιες ανάγκες. Διμερείς τέτοιες συμφωνίες μπορούν κομμένα και ραμμένα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιτόπου και έχουμε τις καλύτερες εμπειρίες που έχουμε συλλέξει με μια τέτοια προσέγγιση για τους ελέγχους. Η πρόταση στο άρθρο 9 εμπεριέχει ρυθμίσεις που υπό το πρίσμα της πρακτικής εφαρμογής δεν συνεισφέρουν για την βελτίωση της υλοποίησης της ε, συμμόρφωσης σε σχέση με την απόσπαση. Οι αρχές θα πρέπει να έχουν επαρκή μέσα στη διάθεσή τους ώστε η τήρηση των ελάχιστων όρων απασχόληση να μπορούν να, ελέγχονται, να ελέγχεται απο, αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα να μπορεί να απαιτείται να υποβάλουν οι επιχειρήσει στοιχεία, έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία θα διασφαλίζεται η καταβολή του ελάχιστου μισθού. Το θέμα, ποια τέτοια έγγραφα είναι αναγκαία για τέτοιου είδους ελέγχους, αναπερίπτωση διαφοροποιείται. Εδώ έχουμε και τις στρατηγικές που διαφοροποιούνται για την παράκαμψη και αποφυγή συμμόρφωσης. Γι' αυτό στη Γερμανία έχουμε διαρκώς μετεξελίξει και προσαρμόσει τις ανάγκες. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της πρότασης, μόνο συγκεκριμένες τέτοιες υποχρεώσεις ε, μπορούν να ε, θεωρούνται δεδομένες. Έτσι τα κράτη-μέλη δεν θα είχαν πλέον δυνατότητα να ανταποκριθούν στις επίκαιρες ε, αλλαγές και προσαρμογές. Εδώ έχουμε τα θέματα του ανοιχτού ή κλειστού πίνακα σε σχέση με το άρθρο 9 για να μπορούν να συμπληρωθούν τέτοιου είδους ελεγκτικά μέτρα εκ νέου, πρέπει τα κράτη-μέλη σε περίπτωση κλειστού καταλόγου να αλλάξουν το πλαίσιο εφαρμογής ώστε να εισαχθεί ένα νέο πλαίσιο υλοποίηση για τα κράτη-μέλη. Έτσι θα μπορούσε με μεγάλη καθυστέρηση να υπάρχει αντίδραση και αυτό θα οδηγούσε σε περιορισμό αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Εμείς πιστεύουμε ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι διατυπωμένα στη γλώσσα του κράτους υποδοχής γιατί διαφορετικά θα πρέπει οι υπάλληλοι να είναι σε θέση να κατέχουν όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό. Στο αντίστοιχο άρθρο προβλέπεται ότι μόνο κάποια συγκεκριμένα έγγραφα θα πρέπει να μπορούν να μεταφραστούν και αυτά όταν δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο εύρος από πλευρά κειμένων. Η δυνατότητα κατάχρηση ε, τέτοιων ε, ρητρών ε, με βάση ιδιαίτερα εκτενή κείμενα είναι δεδομένη. Παραμένει επίσης και το θέμα της, του περιορισμού μετάφρασης ε, <clears throat> σε σχέση με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Περαιτέρω δεν είναι σαφές σε ποιο εύρος θα πρέπει έντυπα και έγγραφα να παραμένουν αποδεκτά σε σχέση με την απόσπαση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακριβείς όροι της απόσπασης. Διαφορετικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί το δίκαιο για τους αποσπωμένους εργαζομένους αποτελεσματικά. Αντιπαραγωγικό θεωρώ ότι είναι και ε, εκείνο το οποίο αναφέρεται στην αρχή όσον αφορά το σκεπτικό 16. Σύμφωνα με αυτό, έλεγχοι θα είναι τότε μόνο εφικτοί αν η ε, ενημέρωση και τα στοιχεία δεν θα μπορούν μέσα σε μια εύλογη προθεσμία να έχουν υποβληθεί από τα κράτη ε, που αποσπούν εργαζομένους. Ιδιαίτερα σε σχέση με ελέγχους ε, επιχειρήσεων θα βελτιωνότανε το πλαίσιο αυτό αν κάποιες επιχειρήσεις δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους βλέπουμε ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό και θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτόπου ελέγχου. Χώρες όπως η Γερμανία που ε, έχουν δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα κατά του του ανταγωνισμού θα πρέπει να στερηθούν αυτές τις δυνατότητες και να δούμε ποια τεράστια προβλήματα δημιουργούνται όταν δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί βλέπουμε ότι υπάρχει μ, επιμερισμός εργασίας σε ένα εργοτάξιο διαφορετικές επιχειρήσεις με διαφορετικούς εργαζόμενους που έχουν αποσπαστεί από διαφορετικά κράτη-μέλη δραστηριοποιούνται. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ισοπεδωτικά να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα με διάφορους περιορισμούς. Τι θα γίνεται, θα διακόπτεται ο έλεγχος ε, όταν, ε, όταν ξαφνικά διαπιστώνεται ύπαρξη κάποιων επιχειρήσεων από ε, κάποια άλλα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να διασφαλίζουμε τα πλαίσια ελέγχου εγώ πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο πρέπει να τροποποιείται σε σημαντικό βαθμό και να προσαρμόζεται ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα πρέπει στο κράτος υποδοχής ε, να δρούμε αποτελεσματικά στους ελέγχους. Οι ελεγκτικές αρχές πρέπει να έχουν επαρκή μέσα στη διάθεσή τους ώστε να μπορούν να ελέγξουν την, το σεβασμό των ελάχιστων αυτών προδιαγραφών υπέρ των εργαζομένων. Θα πρέπει να μπορούν να απαιτήσουν τη διάθεση τέτοιων εγγράφων από τις επιχειρήσεις στη γλώσσα του κράτους υποδοχής. Διαφορετικά είναι αναποτελεσματικός ένας τέτοιος έλεγχος. Η αναλογικότητα μεταξύ κράτους αποστολής και κράτους υποδοχής πρέπει να διασφαλίζεται. Οι έλεγχοι πρέπει καταρχήν επιτόπου να διεξάγονται. Επιτόπου εκεί όπου εργάζονται οι αποσπόμενοι εργαζόμενοι. Θα πρέπει το κράτος το οποίο ασκεί αυτούς τους ελέγχους να είναι ελεύθερο στη διακριτική ευχέρεια αυτών των ελέγχων. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο σαφή και εμπεριστατωμένη ε, άποψη που μας εκθέσατε και γιατί σεβαστήκατε ακριβώς τα 10 λεπτά που είχατε στη διάθεσή σας. Ο κύριος Μαγιόρ έχει τον λόγο τώρα. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, πρακτικές παρατηρήσεις, ε, γιατί καταρχάς εμείς δεν είμαστε ένας οργανισμός ελέγχου, αλλά βλέπουμε τα πράγματα από την ε, σκοπιά των ε, εργαζομένων, των, ε, της εργασίας, του τομέα εργασίας. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα με την οδηγία αυτή δεν θα είναι καλά, θα δημιουργηθεί ένα κάποιο χάος. Ούτως ή άλλως έχουμε και μια οδηγία από το 2004 που αφορά την απόσπαση ε, εκεί εμπεριέχεται ένας ορισμός ε, ο οποίος επαναλαμβάνεται Έχουμε ένα δεύτερο ε, ορισμό για τον αποσπασμένο εργαζόμενο. Ας πούμε ότι έχουμε έναν εργαζόμενο που εργάζεται σε μια μικρή επιχείρηση στην Κρακοβία και πριν αποσπάσει έναν εργαζόμενο του, απευθύνεται στον Οργανισμό Κοινωνικής Απασχόλησης στην Πολωνία και ρωτάει αν γίνεται σεβαστή η κοινωνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λένε ότι όντως είναι όλα, η απάντηση είναι καταφατική και αποσπά τον εργαζόμενο στην Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Και μετά έχουμε έναν Γάλλο επιθεωρητή, ο οποίος θα πρέπει να ε, εξετάσει κατά πόσον γίνεται σεβαστό το άρθρο 3 όσον αφορά την απόσπαση. Και να ξέρετε ότι μιλάμε ε, ότι συχνά συμβαίνουν τέτοιου είδους περιπτώσεις και να έχετε στο μυαλό σας ότι μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις, όχι για μεγάλες επιχειρήσεις. προσπαθούν να σεβαστούν τους κανόνες, θεωρούν ότι τους σέβονται, προχωρούν στην απόσπαση και μετά ελέγχονται για τα κατά πόσον ο δεύτερος ορισμός ε, για, την, για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, ορισμός του άρθρου 3 γίνεται σεβασμός. Φοβάμαι επομένω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και απευθύνομαι ε, στους συγγραφείς, στους εμπνευστές αυτής της ε, ε, οδηγίας. Εάν, ας πούμε, οι αρχές στην Πολωνία λένε ότι όλα είναι εντάξει και ο Γάλλος επιθεωρητής πει όχι, αυτό δεν είναι απόσπαση. Αυτός ο, ο, ο, άνθρωπος έχει έρθει παράνομα εδώ. Είναι παράνομη η απόσπαση. Είναι πρακτικό το πρόβλημα αυτό. Και υπάρχει ορισμός του 883 του 2004 και λέει ότι η χώρα προέλευσης είναι υπεύθυνη. Ο δεύτερος ορισμός όμως του άρθρου 3 λέει ότι το δικαστήριο στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Σουηδία τέλος πάντων θα είναι το κατάλληλο δικαστήριο που θα κρίνει. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι φοβάμαι πραγματικά ότι θα έχουμε δίκες ε, που θα κρατάνε χρόνια ολόκληρα και ε, καταστάσεις ε, ιδιαίτερα περίπλοκες που δεν θα μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Κάτι άλλο, το άρθρο 9. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να αποθηκεύονται έγγραφα. Στον 21ο αιώνα να στέλνουν, που στέλνουμε τα έντυπα με email μέσα δευτερόλεπτα, μπορούμε να, τους, ε, να τα στείλουμε τα έγγραφα μήνες πριν. Εγώ πήρα μία την πρόσκληση, μετά επισκέφθηκα τις, ε, γραμμα... τις γερμανικές τελωνιακές αρχές και η τελωνιακή της Γερμανίας μου είπαν να, μου δείξουν πού αποθηκεύουν τα έντυπα. Και είπα ότι θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εδώ και να πάρω τα έγγραφα και να τα φέρω. Μίλησα με τον υπεύθυνο της επιχείρησης, ε, πέντε μέρες κράτησε αυτή η διαδικασία και μετά το γεύμα, μετά το, ε, τη συνεδρίαση θα, που θα πάμε στο γεύμα και εγώ θα συναντήσω Βέλγους ε, εκπροσώπους ε, ελεγκτές, ε, επιθεωρητές εργασίας και ε, που ελέγχει διάφορες εταιρείε, επιχειρήσεις, ξένες κτλ. Και αν ο Βέλγος επιθεωρητής έχει κάποια, κάποιες απορίες, κάποια προβλήματα και αν γίνει διασταυρούμενη, αν θέλετε, αν γίνει μια συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, θα ζητήσουν κάποια έγγραφα, όμως μιλάμε για επικοινωνία του 21ου αιώνα. Μπορεί να ανταλλαχθούν αυτές οι πληροφορίες άμεσα. Δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε ε, ε, μια υποχρέωση αποθήκευσης εγγράφων και εντύπων. Όταν μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία είναι παρούσα, ας πούμε μικρή επιχείρηση που είναι παρούσα σε 4-5 σε 4-5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλουμε ε, την υποχρέωση σε αυτή την εταιρεία να, έχει, να νοικιάσει γραφεία στις 4 αυτές οι 5 χώρες. Αυτό είναι τεράστιο διοικητικό κόστος. Τώρα και κάτι άλλο. Οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με τα συνδικάτα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ανάγκη επιβάλλει κι άλλο ένα κόστος. Αν δεν κάνω λάθος, δημιουργείται και μια νέα θέση απασχόλησης, έναν διαπραγματευτή δηλαδή. Ας πούμε ότι έχουμε μια, μια αυτή την επιχείρηση, την μικρή επιχείρηση στην Κρακοβία που είναι παρούσα σε 4-5 χώρε. Αυτό τι σημαίνει. Η εταιρεία αυτή θα πρέπει να έχει έναν διαπραγματευτή, έναν επίσημο εκπρόσωπο ο οποίο θα διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα των χωρών αυτών. Τώρα και σε ένα άλλο θέμα κοινή ευθύνη. Αναφερθήκατε στο, στο άρθρο 12 που αναφέρεστε σε όλη την αλυσίδα των εργολάβων και ένας υπεργολάβος γίνεται, ε, επιλέγεται. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε πολύ για την κοινή ευθύνη, διότι πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα επιβάλλει διοικητικό και νομικό χάος το άρθρο 3, πρόεδρε, ε, δημιουργεί πρόβλημα. Αναφερθήκατε στον ορισμό του, του αποσπασμένου εργαζόμενου και μιλήσατε για το άρθρο που αφορά την καταστρατήγηση. Καταστρατήγηση και κατάχρηση του νόμου. Η κυρία Τούρονεν είπε ότι η οδηγία 96-71 δεν λειτουργεί σωστά. Να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συνεργασία, μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές και θα πρέπει η εργατική νομοθεσία σε όλες τις χώρες να είναι σαφής να υπάρχει στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μην έχουμε ε, έτσι ώστε να μην, έχουμε, ε, να μην δυσκολευόμαστε μάλλον να ενημερωνόμαστε άμεσα για το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για τη σαφήνεια και την διαφάνεια των παρατηρήσεών σας. Θα δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά στη συνέχεια. Ο κύριος Γιόνσεν τώρα από τα, ε, τα συνδικάτα της Σουηδίας παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την κοινοβουλευτική σα επιτροπή. Πρέπει να δείξετε κατανόηση. Έχω προετοιμάσει στα αγγλικά αυτόν τον λόγο και θα ε, ήθελα να δείξετε την κατανόηση γι' αυτό. Η απόσπαση εργαζομένων ε, έχουν, βρίσκεται στο επίκεντρο από την ομολογία για την υπόθεση Λαβάλ. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανεργία και τις μεγάλες διαφορές μισθολογικές μεταξύ των κρατών μελών και αυτό φάνηκε ότι είναι ένα τοξικό περιβάλλον πολύ προβληματικό και βλέπουμε ότι αποκαλύφθηκαν προστριβές και προβλήματα όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν ξέρω κατά να έχετε εξοικειωθεί με την ομολογία Ναβάλ, αλλά για την ερμηνεία τη απόσπαση εργαζομένων υπήρξε η θεμελίωση κάποιων αρχών για τη μισθολογική, το μισθολογικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Κάποια όμω ερωτήματα και θέματα τίθενται και κάποια από αυτά είναι ποιο είναι ο συσχετισμό όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική διάσταση και συνιστόσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μια νέα ισορροπία μπορεί να εξευρεθεί. Υπάρχει απορρίθμιση στην Ευρώπη με αυτό το μέσο. Ποιο είναι το εύρο ε, τη ευρωπαϊκή νομοθεσία απεριόριστα καθορίζονται κάποια δικαιώματα εργαζομένων. Ποιο είναι το εύρο ε, για τα μέτρα που θα ισχύουν από τα κράτη-μέλη. Πώ μπορεί ένα ελάχιστο χαρακτήρα για την οδηγία αυτή η απόσπαση εργαζομένων, πώ αυτό μπορεί να αποκατασταθεί και πώ αυτά τα συστήματα, αυτά τα πλαίσια μπορούν να γίνονται σεβαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά, πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάτι θα έχει να προσφέρει υπέρ των εργαζομένων τη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι ο κινητήρα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενωμένη στην πολυμορφία. Να μην επιδεινωθούν τα πράγματα, αλλά να γίνουν πραγματικότητα υπό αυτό το πρίσμα. Η προοπτική των συνδικάτων είναι σχετικά απλή. Όταν βρίσκεσαι στη Ρώμη, να φέρεσαι όπω οι Ρωμαίοι. Δηλαδή, ίση μεταχείριση αποσπόμενων εργαζομένων και σαφείς κανόνε και κανονισμοί όσον αφορά τη χώρα υποδοχή. Αυτά ήταν τα σκεπτικά σε σχέση με την απόσπαση. Οι εργαζόμενοι πρέπει με ίσο τρόπο να, και ισοδίκαιο τρόπο να αντιμετωπίζονται όσον αφορά το πλαίσιο των δικαιωμάτων τους τα ε, σουηδικά συνδικάτα και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα απέτησαν δύο αρχές από τους νομοθέτες μετά από την νομολογία Λαβάλ. Πρώτον, την έγκριση ενός ε, πρωτοκόλου, δηλαδή μια προσαρμογή της συνθήκης, με άλλα λόγια. Και δεύτερον, την ρύθμιση της οδηγίας για την απόσπαση ε, των, δικαιωμα... των εργαζομένων όσον αφορά τα, τα δικαιώματά τους. Ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο σε σχέση με την διάρκεια και την οδηγία απόσπασης. <coughs> εδώ υπάρχει, ας το πω έτσι, η ίσονος ε, ε, διαδικασία, η ίσονος διάστασης ε, ε, εφαρμογή. Και τώρα έχουμε τα προβλήματα της οδηγίας αυτής. Είναι πολύ εύκολο υπό το πρίσμα των συνδικάτων να πει κανείς ότι απογοητευόμαστε υπό το πρίσμα των τόσων λίγων που έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποκατασταθούν τα πλαίσια μέσα από την ομολογία Λαβάλ. Όμως κατανοούμε, δείχνουμε κατανόηση για το ότι είχε πολλά εμπόδια να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δράση και δραστηριοποίησή τη σεβόμενοι τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξευρίσκοντας συμβιβασμούς μεταξύ των κρατών μελών ε, εκεί όπου υπάρχουν και θεσμικές ε, και μισθολογικές και άλλες διαφορές και ταυτόχρονα σεβόμενοι τα αιτήματα των συνδικάτων. Είναι ένα δύσκολο να επιτευχθεί στο, στις απαιτήσει του εγχείρημα αυτό. Τούτων λεχθέντων όμως εκ προημίου θα παρουσιάσω το γενικότερο πλαίσιο όλων αυτών. Να πω δύο λόγια για την προτινόμενη οδηγία συμμόρφωσης και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ στο κάτω-κάτω. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή η πρόταση παρουσιάστηκε με ένα πολιτικό στόχο της διασφάλισης ε, και δικαιωμάτων και διευκόλυνσης ε, της ε, απόσπασης εργαζομένων. Όσον αφορά και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Διασφαλίζονται κάποιες αρχές, δεν θα είναι δυνατόν όλα τα στοιχεία αυτά να τα σχολιάσω, κάποια από αυτά θα μπορέσω να σχολιάσω μόνο φυσικά μπορούμε στη συνέχεια να τα συζητήσουμε πιο εξειδικευμένα όταν θα έρθει η ώρα ερωτήσεων και παρεμβάσεων. ξεκινώντα έλεγχος δημοσίων αρχών. Αυτό είναι το σημείο εκκίνηση για την προτινόμενη οδηγία εφαρμογής. Αφε αυτού είναι κάτι προβληματικό, λέμε εμείς, υπό το πρίσμα των Σουηδικών και γενικότερα Σκανδιναβικών Συνδικάτων. Η πρόταση, θα έλεγα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πρότυπα εργασιακής αγοράς που βρίσκονται στη Ρινανία για παράδειγμα ε, μέσα στα πλαίσια Γερμανίας, ας το πω έτσι, Γαλλογερμανίας. Αυτή αυτό είναι το πνευματικό πλαίσιο με το οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα για να κατανοήσουμε τα στοιχεία αυτής της πρότασης. Κάποια από αυτά τα στοιχεία θα είναι δύσκολο να συμβιβαστούν με άλλα πρότυπα αγορών με την αυτοδέσμευση και αυτοπιθαρχία των εμπλεκόμενων, δηλαδή των κοινωνικών εταίρων όπως τους αποκαλούμε. Όμως ο πιο σημαντικός όρος είναι η μισθολογική όρη η αμοιβή, οι αμοιβή δηλαδή και η όρια απασχόλησης που είναι σημαντικότατα στοιχεία. Το άρθρο 9 στοχεύει στο να περιορίσει τις διοικητικές απαιτήσει όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου που μπορούν και επιτρέπεται να εισαγάγουν τα κράτη-μέλη. Παρότι πολλά από αυτά τα μέτρα τα καλωσορίζουμε, ανησυχούμε με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κλειστό πίνακα. Για οποιονδήποτε προέρχεται από μια φιλελεύθερη δημοκρατική, ας το πω προσέγγιση, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Η ελευθερία είναι η βασική αρχή υπό την οποία πρέπει να λειτουργεί κανείς και ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα κλειστό τέτοιο κατάλογο. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι στην προσέγγιση μας με έναν ανοιχτό κατάλογο. Διαφορετικά όλα απαγορεύονται και πρέπει εδώ να δούμε όχι μόνο ότι δημιουργούνται προβλήματα διοικητικά αλλά υπάρχουν περιορισμοί και νομικοί και δημιουργούνται περιορισμοί για αποτελεσματικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εισαχθούν ανάλογα με τις ανάγκες επιτόπου και κατά καιρών. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιε θα ήταν οι απαιτήσει για ένα οποιοδήποτε τέτοιο περιβάλλον σε 5, 10 ή ε, περισσότερα χρόνια. Γι' αυτό ένα τέτοιο κατάλογο πρέπει να είναι ανοιχτό και όχι κλειστό. Τα άρθρα 5 και 10 στη συνέχεια αντιμετωπίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες και ελέγχους και επιθεωρήσεις. Τι είδους πληροφορίες μπορεί να είναι διαθέσιμες, πού θα είναι διαθέσιμες όλα αυτά κυμαίνονται και παραλλάσσονται από κράτος σε κράτος. Και όσον αφορά επίσης και τα θέματα και τον ρόλο των επιθεωρήσεων. Όπως προανέφερα, συλλογικέ συμβάσεις και επιθεωρήσεις είναι θέματα των κοινωνικών εταίρων στην Σουηδία συλλογικές συμβάσεις ε, θεωρείται ότι είναι μέσα ιδιωτικού, εργαλεία ιδιωτικού δικαίου. Θέματα μεταξύ δύο εμπλεκομένων συμβαλωμένων μερών που ρυθμίζουν κάποιους τομείς. Κατανοούμε φυσικά την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και από την άλλη πλευρά υπάρχει έργο που έχει αναλυφθεί ώστε να υπάρχουν πλαίσια συμφωνιών για τέτοιου είδους αποσπάσεις, ώστε να αυξάνεται η διαφάνεια σε τέτοιες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά όμως οι απαιτήσει για πρόσβαση σε πληροφορίε πρέπει να διασφαλίζονται με την πλήρη ανεξαρτησία και αυτόνομο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και πρέπει να είναι σεβαστά τα διάφορα συστήματα όσον αφορά τους όρους ε, εργασίας και απασχόλησης και όχι μόνο ένα πρότυπο το οποίο υφίσταται στην Ευρώπη ή ένα άλλο. Και α ολοκληρώσω με το άρθρο 3 σε σχέση με θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες αυτό στοχεύει στο να αποσαφινιστεί το τι είναι η απόσπαση. Θεωρώ ότι είναι καλές αυτές οι προθέσεις. Ωστόσο υπάρχει απουσία συνεκτικότητας και λογικής συνάφειας. Ας α, καταστήσω σαφές με απλό τρόπο τι εννοούμε. Ένας από τους στόχους είναι να αποφύγουμε παράκαμψη και υπονόμευση. Αν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση ως έχει σήμερα στη διατύπωσή της, θα μπορούσε το ακριβώς αντίθετο να επιτύχει και όχι τη συμμόρφωση. Αν υιοθετηθεί, τρεις πιθανές νομικές καταστάσεις θα απέρεαν για την απόσπαση εργαζομένων από επιχειρήσεις που θα πρέπει να, διορίζονται, να καθορίζονται από τα κράτη-μέλη που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσε να ήταν γενικότερα θέματα απόσπασης, γενική απόσπαση ως αποκαλείται, η γενική θετική απόσπαση και μετά ένας τρίτος εναλλακτικό τύπος μη γενικού χαρακτήρα, εκτός δηλαδή του πλαισίου απόσπασης απασχόληση. Αυτές είναι με τυπικό χαρακτήρα οι περιπτώσεις εκείνες σε σχέση με την παράκαμψη που θα μπορούσαν να αναφύονται ενώ ο στόχος της οδηγίας είναι να αποφευθούν τέτοιες παρακάμψεις και η απώλεια λογική συνέφειας έχει συνέπειες όσον αφορά και τα παρεπόμενα. Υπάρχει απόλυτη σιγή ηχθείως για το τι θα συνέβαινε με τέτοιους όρους απόσπασης. Πρέπει να αποσαφηνίζεται ωστόσο ότι εκείνες οι επιχειρήσεις δεν πρέπει κάποιες επιχειρήσεις να είναι οι κερδισμένες έναντι κάποιων άλλων. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση σε σχέση με τις χώρες υποδοχής, οι κανονισμοί των οποίων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όπως είπα υπάρχουν και άλλες ε, περιοχές και άλλα πεδία και τομείς. Δεν θα επισέθω σε όλα αυτά. Ο χρόνος πιέζει και ε, αναλώνεται τώρα, εξαντλείται και για αυτή την θετική πρόταση την οποία καλωσορίζουμε πρέπει να υπάρξουν αποσαφηνήσεις. Έχουμε και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Έχετε πολλά χαρτιά και έντυπα τα έγγραφα τα οποία πρέπει να αναγνώσετε και ολοκληρώνω με αυτή την παρατήρηση. Um, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορείτε να μοιράσετε τις απόψεις σας και νομίζω ότι και η συγγήτρια θα είναι θα τις διαβάσω μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις γιατί μας δώσατε μια σαφή εικόνα και σαφείς εξηγήσει και ε, παρουσιάσατε κάποια βασικά θέματα για τα οποία ενδιαφέρεται και η κυρία του Ρένεν του Ρούνεν, συγγνώμη. Ε, έχουμε ε, μέχρι τις 12 η ώρα κάποιο χρόνο να συζητήσουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές Λοιπόν, έχουμε τους τέσσερις σκιώδεις μαζί μας. Α, και την ε, σκιώδη εισηγήτρια ε, για την ε, επιτροπή, από την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα σας προσθέσω τον κατάλογο. Και μετά έχουμε την κυρία Χέντου που θέλει να πάρει το λόγο και τον κύριο Σβάμπ. Uh, λοιπόν, έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα να δώσω την δυνατότητα στους ε, εμπειρογνώμονές μας να απαντήσουν κιόλας. Επομένως, πάλι στα δύο λεπτά, δεν θέλω να σας περιορίσω, αλλά τέλος πάντων πρέπει να έχουμε και κάποιο διάλογο για να μην τα πιέσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους κοιόδης συγητές. Η κυρία Χάνσλικ θα ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας, όλους τους ειδικού και επαΐοντες. Έχουν συνεισφέρει τα μάλα στις συζητήσεις μας ε, για αυτό το σχέδιο οδηγίας. Όλοι συμφωνούμε και ευελπιστώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το σχέδιο στοχεύει στην διασφάλιση ελάχιστου επίπεδου προστασίας των δικαιωμάτων των ε, αποσπόμενων εργαζομένων. Αφενός αυτό από τη μία πλευρά, αφετέρου από την άλλη πλευρά, στόχος είναι να διευκολύνουμε το έργο των παρόχων υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό το δεύτερο στοιχείο, διότι πιστεύω ότι πρέπει να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο στόχων. Πρέπει να διασφαλιστεί η ισορροπία με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό περίγυρο για θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων υπηρεσιών. Αυτή η ισορροπία είναι σοβαρή υπόθεση. Η σοβαρία μεταξύ ελευθερία παροχή υπηρεσιών αφενό και προστασία ε, ε, εργατικών, εργασιακών δικαιωμάτων των αποσπόμενων εργαζομένων αφετέρου. Βλέπουμε ότι τα θέματα τα οποία αναφέρονται από του ειδικού ε, είναι ανησυχητικά και πρέπει να τύχουν τη προσοχή μα. Έχουμε κριτήρια σε σχέση με το άρθρο 3. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί ο δεσμό και η σχέση μεταξύ σχέση κράτους απόσπασης ε, και επιχείρησης για αποσπόμενους εργαζομένους. Η εισαγωγή τέτοιων κριτηρίων σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αξιολόγηση κάθε φορά ανά περίπτωση. Τίθεται το ερώτημα Ποιο θα υλοποιεί και θα είναι υπεύθυνο για αυτή την αξιολόγηση όσον αφορά για την ε, λήψη αποφάσεων και το θέμα επιβολής προστήμων και κυρώσεων αν κάτι δεν βαίνει καλώς. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Ίσως οι επαΐοντες μπορούν να αναφερθούν οι ειδικοί μας σε αυτά τα θέματα. με ο κοινό επιμερισμός αυτών των ευθυνών μπορεί να διασφαλιστεί όταν έχουμε ε, διάφορες επιλογές όσον αφορά υπεργολάβους και θα πρέπει να υπάρχει η σωστή αξιολόγηση μέσα σε ένα εύλογο πλαίσιο για όσους εμπλέκονται υπεργολάβους και επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει μεμονωμένα κάποιοι να θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι υπό το άρθρο 12 εδάφιο 1 το πώς ε, ένας, ε, ε, θα, κάποιος θα πρέπει να αξιολογεί αυτά τα πράγματα συναρτάται με τον τρόπο της λογοδότησης. Επόμενο ερώτημα. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να εξευρεθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σωστά. Για να ολοκληρώσω θα ήθελα να πω ότι αξίζει, είναι, αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις αλλά μέσα σε ένα αναλογικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο αναλογικό. Κανένας δεν επιθυμεί να αποθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις από την χρήση της, του, της δυνατότητας απόσπασης εργαζομένων. Ταυτόχρονα κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές ε, πιθανές επιπτώσεις για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στην Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους ειδικού μας και ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπαρτ, παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης και τους ε, επαΐοντες, τους ειδικού για τις αξιόλογες πληροφορίες πραγματικά που μας ε, ε, έδωσαν. Θα ήταν ενδιαφέρον αν θα μπορούσαμε αυτά με γραπτή, με έντυπη μορφή να μπορέσουμε να τα αναγνώσουμε διότι θα ήταν πραγματικά κάτι το εποφελές για το έργο μας. Για την ομάδα μου ουσιαστικά ήταν απογοήτευση πρέπει να πω να, η επίτευξη αυτής της οδηγίας μετά από την ομολογία Λαβάλ και άλλων περιπτώσεων που προηγήθηκαν, που κατέδειξαν ότι η οδηγία περί απόσπασης δημιουργεί κάποια κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. Αυτό εξακολουθεί και παραμένει αίτημα της ομάδας μας να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και αυτά τα κενά. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η πρόταση ως έχει είναι ανεπαρκής. Ένα περαιτέρω πρόβλημα το οποίο βλέπουμε ότι αναφύεται παρόλα τα θετικά στοιχεία που υφίστανται είναι ότι υπάρχουν κάποιες επιδεινώσεις που σημειώνονται σήμερα κάποιες οπισθοδρομήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει με τροπολογίες να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα αντισταθμίζοντάς τα με τον πιο θετικό τρόπο. Θα πρέπει να περιοριστώ σε τρία θέματα λόγω χρόνου. Το ένα είναι η βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, σε πληροφόρηση για τους εργαζόμενους. Πρέπει να πω ναι, σωστό και σημαντικό αυτό. Αλλά μόνο με μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο δεν νομίζω ότι επαρκεί να, κάνουμε, να δρούμε με αυτόν τον τρόπο. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, γυναίκες και άνδρες, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ατομικά. Ένα μεγάλο μέρος των αποσπόμενων εργαζομένων εργάζονται στον τομέα των οικοδομών. Και δεν νομίζω ότι πολλοί τέτοιοι οικοδόμοι κυκλοφορούν με λάπτοπ, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ε, iPads και τα λοιπά για να πληροφορηθούν από μια ιστοσελίδα το τι ισχύει για αυτούς. Πρέπει και με άλλα μέσα να εργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε άλλα εργαλεία ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες να φτάσουν σε αυτά τα άτομα, σε αυτούς τους αποσπόμενους εργαζόμενους που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύονται επαρκώς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω στους ειδικού μας. Πώς βλέπετε, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωμα και να βελτιωθεί η κατάσταση των αποσπόμενων εργαζομένων. Άρθρο 7 και εφ' ρυθμίζουν τον ρόλο του κράτους υποδοχής όσον αφορά τα θέματα κρατικής ε, ή διοικητική συνεργασίας. Σωστό και αναγκαίο αυτό. Φυσικά το κράτος υποδοχής εκεί όπου πρέπει να μπορούν να διασφαλίζονται καλύτεροι έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζει αυτούς τους ελέγχους. Το κράτος όμως υποδοχής δεν μπορεί να υλοποιεί εκείνους τους ελέγχους που θα πρέπει να ε, διασφαλίζονται από άλλη πλευρά και πιστεύω ότι κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα μας δείξατε τα οποία πρέπει να επιληθούν για να υπάρξει αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Όχι μόνο το κράτος έδρας αλλά και το κράτος υποδοχής πρέπει να έχουν σαφείς προδιαγραφές για το τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι. Με αυτό πρέπει να προχωρήσουμε ε, ξεκάθαρα με τέτοιες διαφοροποιήσεις ώστε το δίκαιο το οποίο θα διαμορφώνεται σύμφωνα με το κράτος την νομοθεσία του κράτους υποδοχής να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Και σε σχέση με τα στοιχεία, σωστά το είπατε, δεν πρέπει να αφήνετε πόρτα και παράθυρο ανοιχτό για παράκαμψη και αποφυγή για τις διατάξεις που εμείς διαμορφώνουμε και διατυπώνουμε εδώ να αντιστρέφονται ή να ε, στρεβλώνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα ένα πράγμα να αποσαφηνίσω. Εξακολουθώ να μην μπορώ να αντιληφθώ κύριε, πρόβλημα, κύριε Μάιερ το πρόβλημα των επιχειρήσεων, το πρόβλημα των επιχειρηματιών αν δεν εργάζονται σωστά και αποτελεσματικά και αυτό το κάνουν πολλοί επιχειρηματίες δεν θέλω τώρα γενικά όλοι να υποπτευόμαστε τους επιχειρηματίες ότι παρακάμπτουν τον νόμο και είναι παράνομοι. Το αντίθετο, πολλοί από αυτούς οι περισσότεροι είναι νόμιμοι και εργάζονται σωστά. Δεν χρειάζεται να έχουν κανένα φόβο για ελέγχους και επιθεωρήσεις. Εμείς θέλουμε τα μαύρα πρόβατα τα ερήφια μεταξύ των επιχειρηματιών να ταυτοποιούνται, να ανοιχνεύονται και να υφίστανται κυρώσεις ε, και διώξεις. Έτσι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το άρθρο 18-19 του ΙΜΗ. Το σύστημα ΙΜΗ έχει ...τα θεμέλια του όχι στην ε, οδηγία περί απόσπασης, αλλά στην αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων και πτυχίων. Γι' αυτό δεν είναι απόλυτα σαφές για μένα. Μήπως ε, υπερβαρύνουμε το όλο συνολικό αυτό σύστημα τώρα όταν και αν εντάσσουμε στην οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων αυτό το πλαίσιο διότι δεν είχε προβλεφθεί ε, ε, ο σύστημα ε, προώθησης της κρατικής συνεργασίας και ελέγχων. Γι' αυτό με τον εισηγητή θα συνεργαστώ τον κύριο Βίλαν που την έκθεσή του κατά την προηγούμενη εβδομάδα την εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Θα συζητήσω μαζί του για να δούμε είναι συνεκτικό και έχει κάποιο νόημα να κάνουμε αυτό το πράγμα για να μην χρειαστεί να τροποποιηθεί και πάλι αυτό το οποίο εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα για να έχει κάποιο νόημα αυτή η δραστηριότητά μας. Γι' αυτό αυτό το οποίο είπατε το ότι το σύστημα ήμι αφεαυτού δεν επαρκεί είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα και να το εξετάσουμε σε βάθος. Και αν μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα σας θα ήταν πολύ χρήσιμο. Τελευταίο ερώτημα προς τον κύριο Γιόνσον, άμεσα και προσωπικά προς αυτόν, διότι ξέρω ότι στα σκανδιναβικά κράτη το σύστημα είναι διαφορετικό σε σχέση με τα συστήματα των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των συνδικάτων Μπορείτε να εξειδικεύσετε κύριε κάπως περισσότερο πώς βλέπετε εσείς το σύστημα των σκανδιναβικών κρατών και ποια στοιχεία από αυτό το σύστημα είναι απόλυτα αναγκαία. Ευχαριστώ για την απάντησή σας εκ προημίου. Yes, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκέφχαρτ. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με τα θέματα του ΙΜΗ. Διάβασα την τελική συμφωνία και υπάρχει σαφής διάταξη για τις υποχρεώσεις ε, των κρατών μελών. Και υπάρχει και αυτή, αυτό το θέμα των, ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ. Ο κύριος Μποζόη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο και θα ήθελα να, ξεκινήσω, να κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσει, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση. Ούτω ή άλλω ε, είναι πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ε, οι, οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως πληροφορημένοι και να, ε, πλήρως ε, προστατευμένοι και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην ε, αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι η οδηγία αυτή θα οδηγήσει σε μια νομική σαφήνεια, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όλους οι κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα περιπλοκή γιατί αλλιώ η απόσπαση των εργαζομένων θα γίνει μη ελκυστική και αυτό θα υποσκάψει την ε, παροχή των υπηρεσιών. Ε, μία ερώτηση προς τον κύριο Παράμο και θα ήθελα επίσης ε, να ζητήσω από τους και από κάποιον άλλον εμπειρογνώμονα να μου απαντήσει. Για τον κύριο Παράμο η ερώτηση αφορά τους υπεργο... τις υπεργολαβίες. Ίσως να δημιουργηθούν κάποια... κάποιες υπερβολικές και συμπροματικές δαπάνες και η υπεργολαβία να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ο όρος due diligence είναι όρος ο οποίος πρέπει να ερμηνευθεί δεν υπάρχει και εδώ ένας κίνδυνος νομικής ασάφειας. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο μετράει είναι η διοικητική συνεργασία και όλα τα, αυτά τα μέτρα, τα κοινά μέτρα, να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να μην ασχοληθούμε μόνο με την κοινή ευθύνη. Η επόμενη ερώτηση είναι απλή περιέργεια. Δεν, ίσως να μην είναι ρεαλιστικό, αλλά Αναφέρομαι στις προθεσμίες ε, που προβλέπονται από το άρθρο 6 για την αμοιβαία συνεργασία. Δύο εβδομάδες, ε, έξι σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, θα ήθελα να, να ακούσω την άποψη των εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Κύριος Δε Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις γενικές καταρχήν. Εμείς δεν έχουμε κοινωνικό κατόφλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχουμε ελάχιστο μισθό. Δεν υπάρχει μια σύμβαση για την ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση, τίποτα όσον αφορά την ε, σύνταξη, τίποτα όσον αφορά ε, το κατόφλι σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει ένας καλός έλεγχος και να γίνουν σεβαστές οι συμβάσεις στις χώρες όπου δουλεύει κανείς και όπου γίνεται σεβαστή η εργασία. Ε, οι αποσπασμένοι κοστίζουν λιγότερο γενικά, τόσο σε, όσον αφορά τις κοινωνικές φορές και όσο και τους μισθούς ε, σε σχέση με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν έλεγχος διότι υπάρχουν διαφορές και αν δεν γίνεται αυτό τότε ε, εκτρεπόμαστε. Δεν συμπαθώ πολύ την προσέγγιση όσον αφορά τις ε, ε, επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν κάποια δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα Ε, είναι κατοχυρωμένα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την προστασία των εργαζομένων με τις νέες προτάσεις και όχι να προσθέσουμε ε, βάρη στις επιχειρήσεις. Γενικά, εγώ ε, είδα την έκθεση που έχει να κάνει με το δίκτυο στα, στο πλαίσιο της ΙΜΠΕΛ Και όταν βλέπει θέματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, μένει κανείς άναυδος. Διαπιστώνει κανείς υπάρχουν οι, οι υπηρεσίε, οι νομικές, οι οποίες ελέγχουν αν υπάρχουν παραβάσεις σε σχέση με το ποινικό δίκαιο, υπάρχει ένα μέρος ελέγχου όσον αφορά την εργασία, το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο πιο, δίκτυο πιο ευρύ για να μπορέσουν να έχουν μια μεγαλύτερη ισχύ ελέγχου. Έτσι μπορεί κανείς να καταλήξει σε κάποια αποτελέσματα. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο στην υποκείμενη πρόταση. ίσως να είχε η Επιτροπή μια, μια ισοσελίδα κεντρική όπου κανείς κάνει συλλογή όλων αυτών των πληροφοριών. Κεντρικά δηλαδή. Να βλέπει όλα όσα αφοράνε τις υπηρεσίες ελέγχου. Αυτά σαν γενικές παρατηρήσεις όπως σας είπα και περιμένω τις αντιδράσεις των πυρογνωμών. Δεν μιλάμε για λιγότερο έλεγχο αλλά να έχουμε ένα καλύτερο έλεγχο ανάμεσα στις υπηρεσίες ελέγχου. Και φυσικά θα πρέπει ο έλεγχος να είναι πιο αφασιστικός, πιο αποτελεσματικός σε μια, στα πλαίσια μια συνεργασίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now, uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Γιασλοβέτσικα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λυπούμε για την καθυστέρηση. Έπρεπε στην Επιτροπή Απασχόλησης να παραμείνω και στην συνέχεια θα ακούσω φυσικά τις απόψεις σας. Τώρα δυστυχώς όμως μόνο μπορώ να επικεντρωθώ στην παρέμβαση του τελευταίου προσκεκλημένου ειδικού. Παρόλα αυτά θα ήθελα να συνεχίσω αυτή την επαφή έχοντας ακούσει τις παρεμβάσεις και έχοντας παρακολουθήσει τα στοιχεία σας και σε έντυπη, έγγραφη μορφή των παρεμβάσεών σας. Αναφέρθηκε ότι στο άρθρο 3 το πρότυπο το οποίο υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόσπαση εργαζομένων επιτρέπει, όπως αναφέρατε, ε, μια πρακτική αρνητικής απόσπασης εκτός νομικού πλαισίου. Συμφωνώ ότι τα κριτήρια δεν είναι σαφή και έχω μία ερώτηση σε σχέση με αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε έναν αυστηρό κλειστό κατάλογο κριτηρίων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεν θα ήταν καλύτερο αν είχαμε κάποιο είδους ε, κατευθυντήριες γραμμές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως προς σε μια τέτοια κατάσταση, δεδομένης μιας τέτοιας κατάστασης που θα εφαρμοζόταν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός αποσπόμενου εργαζόμενου. Δεν είναι μια ερώτηση που απευθύνω μόνο σε εσά, αλλά απευθύνω αυτό το ερώτημα σε όλους τους ε, ειδικού, σε όλους τους Δεύτερο θέμα, η οδηγία δεν καθορίζει επί ποιο χρονικό διάστημα θα ισχύει η απόσπαση χρονικά. Είναι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπει και ρυθμίζει αυτή τη διάρκεια που θα μπορούσε να είναι διάρκειας μέχρι και 24 μηνών. Και πρέπει να πω ότι είμαι προσωπικά εναντίον του περιορισμού της διάρκειας μια ε, ε, μιας τέτοιας απόσπασης. Αν κάποιος είναι σύμβουλος ε, ε απορρέει το ερώτημα πώς μπορούμε να κρίνουμε τη διάρκεια συμβουλευτικών τέτοιων υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με μια τέτοια απόσπαση εργαζομένου. Και ένα άλλο συναφές θέμα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ε, σε σχέση με συνδικάτα, ενώσεις, συλλόγους, συνδικαλιστικούς και συνδικάτων όσον αφορά τις συλλογικές ε, συμβάσεις. Είπατε ότι στη Σουηδία τέτοιου είδους συμβάσεις μπορούν να υπογράφονται και να συνάπτονται διμερώς και τοπικά και να ισχύουν τοπικά. Έχω ερώτημα σε σχέση με το άρθρο 5. Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τέτοιων συμβάσεων και τους κανόνες και κανονισμούς για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων σε μια τέτοια χώρα έχει κέρια σημασία και οι δύο πλευρές αμφωτέρωθεν, δηλαδή οι εργοδότες αλλά και τα συνδικάτα να είναι εξίσου υπεύθυνοι ως αρμόδιοι για την διασφάλιση από πλευρά συνδικάτων των ελευθεριών ε, των, ε, της ε, σύναψης τέτοιων συμβάσεων, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η ευθύνη παροχής διάθεσης πληροφοριών και στοιχείων για τέτοιου είδους συμβάσεις. Θα έπρεπε στα κράτη-μέλη, πιστεύω, να υπάρχει ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί το όργανο ρύθμισης των υποχρεώσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης και Μόνο τότε θα μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι και να δρούμε υπεύθυνα όταν θα έχει παρασχεθεί μια τέτοια πληροφορία, θα, θα έχει δοθεί και ικανοποιηθεί το πλαίσιο πληροφόρησης και ενημέρωσης, ώστε να υπάρχει ε, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δεν μπορούν να περιοριστούν οι ελευθερίες αυτές. Το προσυπογράφω πλήρως. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να απεμπολούμε τις ευθύνες και την λογοδότηση που πρέπει να διασφαλίζεται. Κάνουμε λόγο για την προστασία ε, των εργαζομένων. Κάνουμε λόγο για το συσχετισμό εργοδοτών και συνδικάτων. Πιστεύω ότι η ενημέρωση και πληροφόρηση πρέπει να στοχεύει στους ε, εργαζόμενους. Ε, και εδώ πολλές φορές έχουμε και γλωσσικά, γλωσσικά θέματα τα οποία αφορώνται. Και θα πρέπει εδώ να δούμε, σε σχέση με την ε, Γερμανία για παράδειγμα, ότι τέτοιου είδους έγγραφα πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αγγλικά. Θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί όχι στα γαλλικά, γιατί όχι στα γερμανικά και στα πολωνικά. Στα αγγλικά επειδή είναι μια γλώσσα την οποία μιλούν οι περισσότεροι και κατανοούν οι περισσότεροι. Και θα ήταν πολύ πιο εύκολο για έναν απλό πολίτη, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, να έχει πρόσβαση και να κατανοήσει τέτοιου είδους έγγραφα στα αγγλικά όταν ε, αφορούν την δική του απασχόληση και να μπορούν σε τέτοια, μια τέτοια μετάφραση να είναι προσπελάσιμα. Με συγχωρείτε ένα τελευταίο θέμα, λυπούμε που μακρηγορώ, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους σας ε, τους ειδικού ε, σε, μια ακρόαση στο, στην αίθουσα 5G2 5G3 διορθώνεται, 5G3 σε ακρόαση τη Επιτροπής Απασχόλησης. Θέλω να σας προσκαλέσω σε αυτήν την ακρόαση. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα είναι στις 3 το απόγευμα, 15.00, στην αίθουσα 5G3. Δύο ορόφους πάνω από αυτόν στον οποίο βρισκόμαστε. Στην Επιτροπή Απασχόλησης που θα διοργανώσει αυτή την ακρόαση. Για το απόγευμα μας είπατε, έτσι, μάλιστα για το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε ω αρμόδια ένα από τα προβλήματα, ένα από τα θέματα που αναφέρατε για την οδηγία αυτή, για την πληροφόρηση των εργαζομένων, να υπάρχει μία θηρίδα, μία αρμόδια αρχή που θα πρέπει να διασφαλίζει αυτή την παροχή πληροφοριών. Πρέπει να το δούμε αυτό υπό του όρου αυτή τη πρόταση, ώστε να μπορεί αυτό να διασφαλιστεί. Αν θέλει κάποιο να διασφαλίσει τέτοιου είδου υπηρεσίε, θα πρέπει αυτά να τα γνωρίζει. Θα ήθελα η κυρία Τούρανεν να διασφαλίσει, να δώσει συνέχεια σε αυτήν την πρόταση. Έχουμε άλλους δύο που ε, θέλουν να παρέμβουν. Δεν έχω δυνατότητα να επεκτείνω περισσότερο τον πίνακα αγορητών. Έχουμε διερμηνήσει ε, με περιορισμένη διάρκεια απασχόλησης. Ε, εσείς και μετά ο κύριος Σβάμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους εισηγητές. Εγώ σας Σιλδημοκράτησα είμαι πολύ ανήσυχη με αυτή την πρόταση. Και έχω μια ερώτηση στο Γιούνσον που εκπροσωπεί τα συνδικάτα στην Σουηδία. Έχουμε, έχουμε την πρόταση Κομισιόν για το άρθρο 9 για τη δυνατότητα των χωρών μελών να κάνουν κάποιους ελέγχους. Αυτό περιορίζεται και αυτό επηρεάζει τους κοινωνικούς εταίρους, το οποίο σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των συνδικάτων ε, να μπορούν να ελέγχουν ναι, μειώνονται και γίνεται πιο δύσκολο να δημιουργήσει κανείς συλλογικέ συμβάσεις. Δημιουργούνται κάποια προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνουν διαπραγματεύσεις. Αυτή, αυτός ο περιορισμός θα έχει αρνητικές υποπτήσεις, θα πλήξει τον σκανδινακό που λέγαμε μοντέλο και θα ήθελα να ξέρω τα συνδικάτα, τα σουηδικά, πώς βλέπουν αυτό το θέμα πώς, ποια νιστάσονται, ποια στάση απέναντι στο άρθρο 9 και αν αυτό μπορεί να αλλάξει. Ε, και τι γίνεται αν λαμβάνουν υπόψη και τη θέση του σουηδικού λεγόμενου μοντέλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιες τοπολογίες από τα σουηδικά συνδικάτα. Μπορείτε να τις δείτε. Είμαι βέβαιος ότι θα ε, πιστεί στην προσοχή κύριος Γιόνσεν στη συνέχεια. Τώρα, στρεφόμενος στους βουλευτές. Θα ήθελα να καλέσω να μπορέσετε να παρέμβετε για δύο λεπτά. Λυπούμε για αυτόν τον περιορισμό. Είναι πολύ σύντομη η δυνατότητα αυτή η παρέμβαση. Θα επανέλθουμε με αυτή τη σειρά. Θα έχουν οι επαίοντες την ευκαιρία να απαντήσουν στα όσα θα αναφερθούν. Ο κύριος Σβάμπ πρώτος, ο τελευταίος αγορητής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσίαση των τεσσάρων συναδέλφων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό συμφωνούμε στην Επιτροπή μας ότι πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και διαφάνειας μέσα σε ένα πλαίσιο ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και πρέπει να πω κυρία Γκέπαντ, επειδή δεν κατανοείτε τις επιχειρήσεις, έχουμε τον συνάδελφο ε, που αυτά τα προβλήματα στα ελβετικά σύνορα τα ανέφερε. Όταν κάποιος έχει ε, καταχωρηθεί ε, νόμιμα και που αναφέρεται ότι δεν μπορεί να αποσπαστεί κάποιος ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μπορώ να κατανοήσω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα σε μια τέτοια επιχείρηση και ότι κάποιοι δεν μπορούν να έχουν κάποια έσοδα ε, ε, κάποιες ημέρες. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο η διαφάνεια πρέπει να διασφαλίζεται. Δεν έχω προς εμάς κάποια ερώτηση, αλλά έχω ερώτηση προς τον κύριο Μάιερ. Γιατί οι ορισμοί σε σχέση με τις δύο οδηγίες ή με τον κανονισμό δεν είναι NEA. Γιατί αυτοί οι ορισμοί δεν είναι NEA ε, Ποιο είναι ο λόγο αυτής τη διαφοράς και διαφοροποίηση, κανεί δεν αμφισβητεί την θεμητότητα ελέγχων και την διεξαγωγή ελέγχων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ίσω τίθεται ε, με αυτή την οδηγία διακοπή δηλαδή κάποια ελεκτική ε, πράξη. Αυτό το ερώτημα έχω ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο, Εντάξει. Καθένα τώρα θα έχει δύο λεπτά για να τοποθετηθεί. Ξεκινάμε με εσά κύριε Πάραμο για να τοποθετηθείτε πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το πώς αξιολογείται πώς αξιολογείται εκείνος ο οποίος θα σταθμίζει την ανάγκη της ε, ε, υλοποίησης σε περίπτωση μιας ε, παραβίασης όσον αφορά ένα αναγκαίο πλαίσιο αλληλεγγύης. Κατά κανόνα θα είναι οι υπηρεσίες επιθεωρήσεων, εκείνες που θα πρέπει να ασχολούνται με τέτοιες παράνομες περιπτώσεις. Είναι δύσκολο σε σχέση με τα Υπουργεία να καθορίζουν ποιες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες εμπλέκονται και ποιες όχι όσον αφορά το σεβασμό τέτοιων διατάξεων. Για το σύστημα ΙΜΗ, αν επαρκεί ή όχι ο σύστημα το ΙΜΗ. Εδώ στην παρέμβαση που έκανα διαφοροποίησα μεταξύ της ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι το σύστημα ΙΜΗ είναι ένα τέλειο εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά απλά πρέπει να δούμε ότι στα θέματα αμοιβαίας αρρωγής, στα οποία υπάρχει ε, συνεργασία, διοικητική συνεργασία που έχει ήδη ξεκινήσει, πρέπει να δώσουμε στο σύστημα ΙΜΗ τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, γιατί δεν πρόκειται μόνο για ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και για ένα βήμα παραπέρα που πρέπει να διασφαλίσουμε. Όσον αφορά με την ευθύνη αλληλεγγύης, όσον αφορά και τις υπεργολαβίες και τις άλλες επιχειρήσεις, Τίθεται το ερώτημα αν αυτό θα είναι επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις ή όχι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα θέμα είναι η νομική επίπτωση που θα μπορούσε να έχει αυτό το σύστημα σε εκείνες τις χώρες που δεν έχουν ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις έναντι εκείνων των κρατών που έχουν νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θα είναι οι ίδιες οι επιπτώσεις φυσικά αυτών των μέτρων. Τούτου λεχθέντος, αν αυτό θα είναι επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις ή όχι, με βάση την πείρα των επιθεωρήσεων εργασίας βλέπουμε με σαφή τρόπο για τους ε, ελέγχους αυτούς ότι δεν είναι οικονομική επιβάρυνση σε καμιά περίπτωση. Είναι επιβάρυνση διαχείρισης, επιβάρυνση ελέγχου. Εκείνο περί του οποίου πρόκειται είναι να υπάρχει έλεγχος ποιοι εργάζονται και πώς ε, σε αυτές τις ε, επιθεωρήσεις για τις υπερ, υπεργολαβίες τέτοιου είδους στοιχεία θα είναι αποτρεπτικά διότι θα αποκλειστούν από την αγορά εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν σέβονται τις διατάξεις και τους κανονισμούς και δεν συμμορφώνονται με αυτούς. Επιπλέον η μεγαλύτερη πειθαρχία και αυστηρότητα θα αντισταθμίζεται με την αναγκαία πειθαρχία και τον αναγκαίο ζήλο που θα επιδεικνύουν οι εμπλεκόμενοι. Με τους σωστούς ελέγχους θα μπορεί λοιπόν να επιμερίζεται το θέμα των ευθυνών. Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορούν να διώκονται οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν αυτές τις αρχές που προέρχονται από άλλες χώρες και που δεν υλοποιούν αυτές τις προδιαγραφές. Υπενθυμίζω και επανέρχομαι στο θέμα θυμπέλες, κυβέλη. Δεν είναι εύκολο να υπάρξουν κυρώσεις διότι δεν υλοποιούνται αυτές οι κυρώσεις και τα πρόστιμα από μια χώρα σε άλλη. Έχουμε χιλιάδες τέτοια πρόστιμα και κυρώσεις που δεν έχουν ε, καμία επίπτωση σε άλλες επιχειρήσεις εκτός Ισπανίας. Και αυτό είναι κάτι το αρνητικό και πρέπει να επανορθωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φον Πρόισεν. Σας ευχαριστώ να επανέλθω στο θέμα του τι είναι έλεγχος ε, και ποιοι έλεγχοι θα γίνονται στο μέλλον. Να απαντήσω καταρχήν λέγοντας ότι πρέπει φυσικά να δούμε το θέμα του 16. Έχουμε ένα θέμα ζήτησης το οποίο πρέπει να θεσπίζεται που στο κράτος ε, προέλευσης για τις επιχειρήσεις του κράτους προέλευσης πρέπει να απαντηθεί. Τήρηση προθεσμιών που στο ε, άρθρο αυτό αναφέρονται σε συνάρτηση με το σύστημα ΙΜΗ. E αν δεν τα καταφέρουμε επιτόπου σε ένα εργοτάξιο να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα και να ελέγξουμε και να δούμε τι γίνεται μεταξύ κράτους αποστολής και κράτους υποδοχής και τι έχει συμφωνηθεί συμβατικά μεταξύ αυτών, τότε θα πρέπει ο έλεγχος αυτός να σταματήσει, να σταματήσει αυτή η δραστηριοποίηση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το αμφισβητήσιμο όσον αφορά την υλοποίηση και επίτευξη των όρων Απασχόληση στο κράτο υποδοχή Στο άρθρο 9 είναι σημαντικό το θέμα του ανοιχτού καταλόγου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κλειστό κατάλογο. Εμεί θα επιθυμούσαμε να είναι ένα ανοιχτό κατάλογος Αυτό. Μια και τακτικά απορρέουν προσαρμογέ και αλλαγέ λόγω τεχνικών όρων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ενταχθεί σε αυτόν τον κατάλογο και πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια πολύ δαπανηρή διαδικασία αν θέλουμε να τροποποιήσουμε και πάλι αυτό τον κατάλογο. Περνάνε δύο-τρία χρόνια όπως είναι αναγκαίο μέχρι επιτόπου να μπορέσουμε στους ελέγχους να προσφέρουμε λύσεις στα νέα προβλήματα. Αυτά είναι θέματα που σε σχέση με τέτοιου είδους ε, ελέγχους ε, πρέπει να τα δούμε διότι δεν είναι δυνατόν η έλεγχη αυτή να είναι αποτελεσματική μέσα σε τέτοια πλαίσια. Τώρα για τα εργοτάξια όσον αφορά τον τομέα των οικοδομών. Είναι κλασικό παράδειγμα αυτό. Υπάρχουν πολύ διαφορετικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε τέτοια πλαίσια. Πολύ δύσκολο θα μπορούσε να δύσκολα θα μπορούσε να διαπιστωθεί από ποιε χώρε προέρχονται όλοι αυτοί οι απασχολούμενοι. Και αυτά να τα πω ότι σε σχέση με τη βοήθεια των συναδέλφων από άλλα κράτη πρέπει να διασφαλιστεί τι συμβαίνει εκεί και μετά να γίνουν οι έλεγχοι. Όλα αυτά είναι πολύ επιβαρημένες διαδικασίες και δίσκαμπτες. Να επανέλθω στο άρθρο 3 που θέλω να το αναφέρω. Έχουμε ένα άρθρο εδώ ενώπιον μας το οποίο ας το πω έτσι την διοικητική συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράκαμψης και της μη συμμόρφωσης πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα και να καταλήξουμε σε ένα αποδεκτό λειτουργικό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα αποδεκτό από όλους όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων. Να το σκεφτούμε καλά δηλαδή σε σχέση με αυτό το άρθρο τι επιθυμούμε να γίνει ακριβώς. Thank ευχαριστώ κύριος Μάιτ. Ευχαριστώ και θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Σβάμπ για τις διαφορές στους ορισμούς για την απόσπαση εργαζομένων γιατί διαφέρουν οι, οι ορισμοί αυτοί και σε σχέση και με την κοινωνική ασφάλιση και αυτά που έχουμε μπροστά μας υπό το άρθρο 3 της τρέχουσας πρότασης. Το πλαίσιο είναι παρόμοιο με μια πρώτη ματιά αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να καταδείξω πού υφίσταται το πρόβλημα το οποίο αναφύεται με βάση αυτά τα οποία εξετάζουμε υπό το 883 υπό το πλαίσιο των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε στο Βέλγιο βελγικά όργανα, στη Γαλλία γαλλικά. Υποθέτουμε ότι αντιμετωπίζουμε θέματα απόσπασης εργαζομένων σε ένα 25% του κύκλου εργασιών σε σχέση με την ε, χώρα υποδοχής. Ισχύει το 25% σε σχέση με το κράτος υποδοχής. Στη δική μου χώρα την Πολωνία έχουμε το 100% για αυτά τα κριτήρια όσον αφορά το 883 και έχουμε και την περίπτωση του Βρότσλαβ όπου ένα περιφερειακό δικαστήριο του Βρότσλαβ σε σχέση με απόφαση που επιβεβαιώθηκε από το εφετείο ότι όταν ισχύουν αυτές οι αρχές για κάποιον Πολωνό έχουμε για περίπτωση της Πολωνίας για παράδειγμα το 7 ή 8% ε, έχουμε τα αντίστοιχα έγγραφα και έντυπα που δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών που απαιτείται να ε, υλοποιείται είναι 50 σε άλλες περιπτώσεις 25% και δίδεται ένα πιστοποιητικό Α1 όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό κύκλου εργασιών. Πήγα στο Βουκουρέστι πρόσφατα. Αυτά που έζησα και βίωσα στο Βουκουρέστι για έξι μήνες, σε έξι μήνες, κανένας επιχειρηματίας που ήθελε να εξαγάγει δεν έπαιρνε αυτό το πιστοποιητικό αν να απεδείκνυε ότι είχε 50% κύκλου εργασίας σε άλλη χώρα υποδοχής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αρχές, διαφορετικές διατάξεις που αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Αυτό ανταποκρίνεται ακριβώς ως κατάσταση στις, ε, στους διαφορετικούς ορισμούς και δημιουργείται χάος μέσα από μια τέτοια κατάσταση. Και θα είχαμε και την περίπτωση της Γερμανίας που θα έπρεπε να αποφασίζει γερμανικό δικαστήριο το τι συμβαίνει, ενώ στην Πολωνία θα ισχύει γερμα... στην πολωνικό δικαστήριο. Δεν έχουν οι επιχειρηματίες φόβο για τέτοιες περιπτώσεις. Ελέγχονται για τέτοιες δράσεις ε, στο εξωτερικό, ακόμα και σε σχέση με τα τελωνία, περί του οποίου πρόκειται είναι οι επιχειρήσεις από την Ανατολική Ευρώπη ή γενικά όσοι δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να μην έχουν επιπρόσθετες ε, υποχρεώσεις που δημιουργούν επιπρόσθετες δαπάνες και επιπρόσθετη επιβάρηση. Μόνο περί αυτού πρόκειται. Και θα ήθελα να αναφέρω και στη συνέχεια κάτι άλλο μετά από αυτή την παρέμβασή μου στα γερμανικά. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την αλλαγή γλωσσών από τα γερμανικά στα πολωνικά. Ας έχουμε μία ρύθμιση. Ας καθορίσουμε στο άρθρο 3 ότι τα θέματα απόσπασης θα αντιμετωπίζονται με τα πρότυπα του Α1 εντύπου. Αυτό ισχύει και ίσχυε στη Γερμανία από το 2004. Αυτή ήταν η πρακτική με την οποία αντιμετώπιζε η Γερμανία και τα οι τελωνιακές αρχές στη Γερμανία αυτά τα θέματα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά από όσα γνωρίζω, αν ισχύει το έντυπο αυτό του Α1, τότε αποδεικνύεται ότι υπάρχει απόσπαση. Ε, ας παραμείνουμε σε ένα τέτοιο ενιαίο πλαίσιο για την απόσπαση. Αυτό καταδεικνύει τώρα το πώς διαφοροποιούνται τα πράγματα ανάλογα με την ομολογία δικαστηρίων. Ε, παρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ για αυτή τη ζωντανή συζήτηση και τη συνεισφορά σας. Και ίσως και το απόγευμα, δύο ρόφους πιο πάνω στην ακρόαση, μπορείτε να ε, συμμετάσχετε. Εσείς κύριε Γιόνσον για τις παρεμβάσεις αυτές μπορείτε γοργά να αντιδράσετε γιατί ο εισηγητή περιμένει τώρα για το επόμενο θέμα και θέλω η κυρία Τουρούνε να μπορέσει στο τέλο να συνοψίσει τι απόψει τη. Να μην ξεχάσουμε τον εισηγητή. Ο κύριο Γιόνσον. Θα είμαι σύντομο γιατί πολλέ ε, απαντήσει μπορούν να δοθούν και μέσω των τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν κάποια ε, σχόλια για το σουηδικό μοντέλο, που είναι το σκανδιναβικό μοντέλο λίγο πολύ, θα δείτε ότι στη Δανία και στη Σουηδία Υπάρχουν ε, ε, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει υποχρέωση για δεσμευτικές συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει μισολογική προστασία κτλ. Στην Σουηδία και στην Δανία έχουμε 600 διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις και όλες αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πραγματικότητες της αγοράς εργασίας γιατί η ανάγκη για την ρύθμιση των μισθών είναι διαφορετική για τους γιατρούς από ότι για τους οικοδόμους παραδείγματος χάρη και οποιοδήποτε ε, ξέρει την αγορά εργασίας θα ε, ξέρει ότι υπάρχουν διαφορετικές υποαγορές. Δηλαδή, ούτω ή άλλω δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί όλοι να είναι πιλότοι, α πούμε. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ε, τώρα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε διαφάνεια όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως σας είπα, έχουμε 600 διαφορετικές ε, συλλογικές συμβάσεις ε, που εξελίσσονται εδώ και 100 χρόνια σε ορισμένε περιπτώσει. Επομένω, δεν είναι εύκολο να τι κάνουμε διαφανεί. Ε, έστω και αν είναι δύσκολο αυτό. Δεν πρόκειται να πω στο κείμενο, σε λεπτομέρειες. Ακούσα, ξέρετε ποιες είναι οι τροπολογίες, ακούσα τις απόψεις μας. Θα είμαι εδώ όλη την μέρα στη διάθεσή σας. Λοιπόν, ευχαριστώ όλοι ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και τους τέσσερις ε, για την ε, παρουσίαση και για τις απαντήσεις που δώσατε, κυρία Τούρουνεν. Α, ε, λίγα λόγια, λίγα λόγια. Ναι, έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά συμφωνώ με κάποιους που είπαν ότι από νομικής πλευράς τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Έχουμε την αρχική οδηγία, μετά έχουμε την ε, οδηγία 883. Μετά έχουμε τις, ε, την προσωρινή απασχόληση. Ε, έχουμε πολλές οδηγίες, είναι ένα patchwork και πρέπει να λειτουργήσει όλο αυτό. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω, σαν απάντηση και στον κύριο Μάιορ, είναι ότι μιλάμε για lex specialis πρέπει να καθορίσουμε εδώ την απόσπαση και εδώ αυτό θα είναι το βασικό κείμενο, διότι το 96 είχαμε ένα πολύ ευρώ ορισμό, ε, ευρύ ορισμό. Από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, δεν θα έχουμε διαφορετικά επίπεδα, απλώς θα διευκρινίσουμε, θα ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε εδώ. Εδώ γίνεται μια εξειδίκευση, αν θέλετε, μια διευκρίνηση του 96. Δεν πρόκειται να δώσω απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Σημείωσα τα πάντα και από τους κοιόδης συζητητές και από τους εμπειρογνώμονες ε, και προσβλέπω στην συνεργασία όλων και εδώ και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι θα πετύχουμε μια ισορροπία ε, όλοι είπαν την άποψή τους, θα την λάβουμε υπόψη μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση όσο έχει τώρα ε, χαρακτηρίζεται από κάποια ανισορροπία και η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί καλά. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και να, ε, για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. έχουμε και εμπειρογνώμονες της Κομισιόν, βέβαια. Green και Φινστρα. Προφανώς ε, θα έχετε την ευκαιρία να μας πείτε την ε, άποψή σας όταν η κυρία Τουρούνεν υποβάλλει την ε, γνωμοδότησή της, γι' αυτό, την έκθεσή της. Γι' αυτό δεν σας δώσαμε το λόγο σήμερα. Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου θα ζητηθεί η έκθεση και 6 Νοεμβρίου η υποβολή, η προθεσμία προβολή των προθεσμιών. Ευχαριστώ και τον Σεμπάστιαν, λέει η κυρία Ρούνιν. Λοιπόν, ε, τελείωσε αυτό το θέμα και όσοι δεν θα ασχοληθούν με το επόμενο, σας παρακαλώ να αποσυρθείτε ησύχως. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα καλωσορίζω τον κύριο Τσαρκόφσκι για την επανεχρησιμοποίηση των πληροφοριών στον δημόσιο τομέα. If Εάν θέλετε να συζητήσετε, μήπως θα μπορούσατε να συνεχίσετε εκτός ευθούσης, σας παρακαλώ. Διότι πρέπει να συνεχίσουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο μέχρι το διάλειμμα. Okay, so could you please, uh, thank you very much. Ευχαριστώ.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 Ε, αυτή η προσέγγιση ακούστηκε ότι μπορεί να είναι ε, δύσκολη, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όσον αφορά τα τέλη υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες τροπολογίες. Τώρα υποστηρίζω επίσης ότι το περιθωριακό κόστος πρέπει να είναι το κόστος το οποίο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο αίτημα. Συμφωνώ επίσης με κάποιες από τις ανησυχίες σας. Ε, βέβαια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να απαιτηθεί ε, περαιτέρω χρηματοδότηση για την ε, εφαρμογή αυτής της οδηγίας και ίσως ε, οι υποδομές, να χρειαστούν υποδομές και πόροι περαιτέρω επενδύσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Προς αναφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πάρα πολλές από τις τροπολογίες σας Είδαμε πώς σχετίζεται η επαναχρησιμοποίηση με την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, συγκεκριμένες τροπολογίες. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Άκουσα τι είπε η κυρία Ρούλε και η κυρία Έγκστρομ. Επίσης, τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπου κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή μία ομάδα αναγνωρίζεται. Πιστεύω ότι το να μιλάμε για προσωποποίηση ίσως να προχωράμε λίγο μακριά. Γιατί είναι και θέμα προστασίας των δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Τέλος πάντων όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας όταν συντάσσουμε τις συμβιβαστικές ε, πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα τα πολιτιστικά ιδρύματα, αυτό συζητήθηκε και στην Πολιτιστική Επιτροπή, Επιτροπή Πολιτισμού, συγγνώμη, και σαν εισηγητής θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ειδικό τρόπο Πάντως η κυρία Φεχέν έχει κάνει κάποιες προτάσεις, τις οποίες θα λάβουμε υπόψη μας. Δύο θέματα ίσονος ε, ε, σημασίας. Ακούστηκαν κάποιες απόψεις για, την, για τα ερευνητικά κέντρα τα οποία πληρώνονται με δημόσιους πόρους. Αυτά εξαιρούνται, αλλά θα πρέπει να το συγκροτήσουμε την Κομισιόν ε, δεν είναι εκπρόσωποι της Κομισιόν εδώ, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα των κατευθυντηρίων γραμμών. Διότι θέλουμε η Κομισιόν να συντάξει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, δεν θέλουμε όμως αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να πάνε λίγο μακριά, δεν θέλουμε να είναι αντιπαραγωγικές, θέλουμε να διευκρινίσουν ορισμένα θέμα και ούτε να, θέματα και όχι να είναι και υποχρεωτικές ούτως ή άλλως, διότι μπορούν ε, οι απόψεις μας όσον αφορά για την, την ψηφιοποίηση να είναι αντιπαραγωγικές. Ε, αυτά είναι θέματα για τα οποία πρέπει να απαντήσει η Κομισιόν για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τις ε, συνεισφορές, για τις συνεισφορές του συναδέλφου. Μου ανοίξετε τα μάτια, οφείλω να ομολογήσω. Κάποιες τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να τις λάβουμε υπόψη μας πλήρως όσον αφορά ας πούμε την Επιτροπή Πολιτισμού και τις ιδιαιτερότητές της ή θα τις λάβουμε υπόψη μας μέσω των νέων συμβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω τον κύριο Σέτενα, ο οποίος είναι πολύ τακτικός επισκέπτης της Επιτροπής μας. Της Επιτροπής μας. Λοιπόν, η κυρία Βάιλερ είναι η πρώτη ε, από τους κοιόδης ηγητές που θα Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη, γιατί ήδη στην πρώτη συζήτηση που είχαμε είπα ότι την προσέγγιση αυτή την βρίσκω σωστή και ότι λίγες τροπολογίες σχετικά θα καταθέσω. Παρ' αυτά, είναι σημαντικό αυτό το θέμα για μένα. Και βρίσκω τροπολογίες από πλευρά συναδέλφου αξιόλογες και τις υποστηρίζουμε. Πάμε ένα βήμα παραπέρα με τις αρχές αυτές. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίζουν τα ίδια. Δεν χρειαζόμαστε ξεχωριστές αρχές. Οι ίδιοι πόροι των κρατών μελών επαρκούν. Αλλά αν το δια, διατυπώσετε έτσι ότι αποκεντρωμένα θα αποφασίζετε αυτό, θα μπορούσα να το δεχτώ. Οι διαθέσιμοι πόροι σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο στη Γερμανία, επαρκούν για να γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ σε διετής περιόδους να έχουμε σύνταξη έκθεσης. Να δούμε και τις κατευθυντήριες γραμμές που εντάσσονται εδώ σε αυτό το πλαίσιο και ο, ετήσ, εισηγητής ήθελε ετήσια να υποβάλλεται τέτοια έκθεση. Αν κάθε δύο χρόνια όμως μας υποβάλλεται τέτοια έκθεση θα μπορούσε να είναι πιο ουσιώδης. Για μια πρώτη αξιολόγηση μπορούμε να δούμε αν είναι ε, ικανές αυτές οι διατάξεις ή όχι. Μπορούμε σε σχέση με μια τέτοια έκθεση σε διετή περίοδο να την έχουμε για να δούμε τα θέματα μεταρρύθμισης και για την 38 από πλευρά Ρούλε θα μπορούσα να την υποστηρίξω. Ένα πράγμα τέλος, τέλος θέλω να πω. Μια παρατήρηση να κάνω στο τέλος. Θα έπρεπε φυσικά πρέπει τα, τα κόστη να τα κρατούμε χαμηλά και προσιτά. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουν τα όρια αυτά τα κόστη. Δεν πρέπει όμως αυτό να είναι ένα κενό, ένα χάσμα να έχουν υπερβολικό, υπερβολικές δαπάνες ε, οι κοινότητες και με αυτό να έχουν ένα παράθυρο για την υπεκφυγή ή αποφυγή. Είναι το μόνο σημείο αυτό. Για το 39 έχω κάποια τέτοια μικροπροβλήματα. Για τα άλλα βρίσκω ότι είναι μια καλή έκθεση και την δέχομαι. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω σαφώς τρία σημεία από πλευράς ε, της ε, διατύπωσης του συντάκτη ή του εισηγητή. Θα πρέπει αυτά τα έντυπα να μπορούν να ε, τα διαβάζουν μηχανές με αυτόματη ανάγνωση. Υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση όσον αφορά την ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει σε σχέση με τους πόρους, όπως είπατε κυρία, εσείς κυρία Βάιλερ, να πούμε ότι οι πόροι επαρκούν πλήρως και έτσι αυτό το δεχόμαστε. Τώρα για την έκθεση που προτείνεται τήσια να συντάσσεται, εμείς θα λέγαμε και κάθε τρία χρόνια μπορεί να υποβάλλεται. Τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένα να ψηφιοποιούν τέτοιου είδους στοιχεία ή τέτοιου είδους έγγραφα. Πρέπει κατά τη δική τους ελεύθερη διακριτική, ε, ελεύθερη διάκριση να μπορούν να αποφασίζουν τι θα κάνουν. Αυτή είναι μια μικρή διαφοροποίηση. Αν θα συμβαίνει και όταν θα συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχουν ενιαίε προδιαγραφές μάλιστα ή ένα ενιαίο πλαίσιο, ένα ενιαίο ε, έντυπο στις ε, διαστάσεις του ώστε να μην υπάρχει ε, κάποια παρέκκληση. Αυτό είναι στις ε, τροπολογίες 18, 19, 21 ε, όμως ε, δεν πρέπει να υπάρχει πρόσθετη δαπάνη που θα απαιτείται. Κατ' εξαίρεση μπορεί να ξεπερνάμε αυτόν τον κανόνα και έτσι ευθυγραμμίζω με τη, με τη δική σας παρέμβαση, όμως είσαστε εναντίον του να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις με αρχεία, βιβλιοθήκες, τέτοιου είδους εξαιρέσεις πρέπει να τεκμηριώνονται, αλλά πρέπει να μπορούν να είναι εφικτές όσον αφορά τις αντίστοιχες τροπολογίες, όσον αφορά την έρευνα. Θα έπρεπε την αρχή της επικουρικότητας να τηρούμε. Στο πλαίσιο, έρευνας, στο πλαίσιο ε, για την έρευνα έχουμε σαφείς κανονισμούς για τη δημοσιοποίηση για παράδειγμα. Όπου κάποιο τέτοιο αγαθό ε, προβλέπεται θα πρέπει να υπάρχει και η δημοσιοποίησή του. Για τη χρηματοδότηση της έρευνας ε, απαιτείται από τους ερευνητές που χρησιμοποιούν τέτοια κονδύλια να αποδεικνύουν το τι κάνουν με αυτά τα χρήματα των κονδυλίων. Δηλαδή όσα αφορά Όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, δέσμευση για δημοσιοποίηση, ότι γίνεται στο εθνικό επίπεδο είναι στη δική τους διακριτική ευχέρεια. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Ρούλε. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Όμως ένα σημείο θέλω να αποσαφηνίσω όταν είπε στην αρχή ότι πρόκειται για την πρόσβαση των πολιτών. Δεν πρόκειται για αυτό. Πρόκειται για την εμπορική χρήση δημόσιων προδιαγραφών και στοιχείων. Δηλαδή τι κάνουν με αυτά τα στοιχεία εκείνοι που τα χρησιμοποιούν εμπορικά. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Βάιλερ, ωραίο ακούγεται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση, το υποστηρίζω αυτό. Αν δούμε όμως την πραγματικότητα, την πραγματική εφαρμογή, ε, γίνονται διάφορα πράγματα, τόμ-τόμ ε, ε, και άλλες περιπτώσεις Εκείνοι έχουν το μεγαλύτερο συμφέρον για τέτοια πρόσβαση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τέτοια στοιχεία και να τα εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλουν να έχουν κάποια κέρδη τα οποία σημειώνουν με αυτή την εμπορική ε, εκμετάλλευση. Και η δημόσια αρχή αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζει, οι κρατικές αρχές αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Έχουμε κράτη-μέλη με μεγάλη υπερχρέωση Βιβλιοθήκες κλείνουν σε πολλά κράτη-μέλη και είναι πραγματικά εύθετο ο κρατικός τομέας να απο ε, τα κονδύλια των φορολογουμένων και να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με την ε, εμπορική διάθεση τέτοιων στοιχείων και εκείνοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια στοιχεία εμπορικά πρέπει να συνεισφέρουν και να πληρώνουν τέλη και εισφορές. Δεν είναι δυνατόν τα στοιχεία τα οποία με τα χρήματα φορολογουμένων έχουν χρηματοδοτηθεί να διατίθενται σε κάποιους που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά δωρεάν ειλικρινά αυτό το πρόβλημα σχετικά αργά το αναγνώρισα, το ομολογώ αυτό και είχα κινήσει από το ότι επρόκειτο σε πρώτη γραμμή για πρόσβαση πολιτών, γυναικών και ανδρών. Πρέπει όμως να πω ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροφής και αν κάποιος αναγνώστης έχει κάποια πίεση με την οποία εργάζεται δεν μπορεί να την ε, αντιληφθεί στο πλήρες εύρος της. Γι' αυτό παρακαλώ να υποστηρίξετε κατεπηγόντως τις ε, τροπολογίες της κυρίας Φαχάν γιατί είναι οι καλύτερες που έχουν κατατέθει. Ευχαριστώ. Okay, Σε ευχαριστώ κυρία Φεχάνη. Επόμενη, παρακαλώ, σύντομο το σχόλιο σας. Σα ευχαριστώ πολύ. Ήμουν εγώ η εισηγήτρια στην Επιτροπή Πολιτισμικών Υποθέσεων για αυτό το χαρτοφυλάκιο Πράγμα το οποίο επεξηγεί και γιατί είχα καταθέσει περισσότερες τροπολογίες από πλευρά μου για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι σαφές πλέον ότι εδώ δεν πρόκειται για ρύθμιση για την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πολίτες. Πρόκειται για την ρύθμιση κριτηρίων υπό ποιου όρους θα πρέπει να δημοσιοποιούνται κάποια στοιχεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από κάποιους. Και εδώ σε πρώτη γραμμή πρόκειται για την εμπορική χρήση αυτών των στοιχείων όχι για εκείνη την οποία ως ιδιώτης εγώ θέλω να έχω για τη χρήση τους. Δεν πρόκειται όμως για αυτό το πεδίο εφαρμογής, αλλά για την εμπορική χρήση. Όχι για πρόσβαση δηλαδή για τους πολίτες, αλλά για την εμπορική εκμετάλλευση από κάποιους. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχει όμως και ένα τεράστιο κοινωνικό δυναμικό εδώ, όταν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί περαιτέρω τέτοιου είδους στοιχεία. Έθεσε η κυρία Ρούιλε το ερώτημα. Ποιο είναι εκείνος ο οποίος αποκομίζει τα κυριότερα κέρδη από τέτοιου είδου στοιχεία και τι γίνεται με τις καινοτόμες υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία βέβαια. Και πρόσφατα στην Αμερική είχαμε κάποια inputs, κάποιες προτάσεις, κάποιες ε, ε, πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και είδαμε πολλές επιχειρήσεις ε, δημιουργήθηκαν που ασχολούνται με την εκμετάλλευση τέτοιων στοιχείων. Πρέπει να δούμε όμως ότι σε σχέση με τις ε, επιχειρήσεις μας ε, πρέπει να ε, επικεντρωνόμαστε στις μικρομεσαίες και στις μικρές. Είναι ένα από τα κυριότερα σημεία της οδηγίας. Η διεύρυνση της οδηγίας αυτής στον πολιτισμικό τομέα που μέχρι σήμερα εξαιρείτο. Πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Μέσα σε τέτοια εγχειρήματα ψηφιοποίησης είναι ανάγκη να έχουμε την υποστήριξη των ιδιωτών δεν είναι δυνατόν διαφορετικά να ενεργοποιηθούμε για την ψηφιοποίηση. Δεν γίνεται χωρίς κόστος και χωρίς δαπάνες μια τέτοια ψηφιοποίηση. Γι' αυτό είναι σημαντικό σε αυτόν τον τομέα του πολιτισμού να προβλεφθούν κάποιες εξαιρέσεις, να είναι δυνατόν να υπάρχουν αποκλειστικού είδους συμβάσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τέτοιες ε, δραστηριότητες. Γι' αυτό είχα καταθέσει τέτοιες τροπολογίες προς όφελος της ε, προώθησης της ψηφιοποίησης ε, πολιτισμικών αγαθών. Και θα πρέπει να υπάρχει τέτοια δυνατότητα για να μπορούμε να δράσουμε έτσι. Έχω αρκετές πολλές τροπολογίες που διατύπωσα, διότι στο ένα ή άλλο σημείο υπάρχουν ανάγκες αποσαφήνισης, πιστεύω επειδή η οδηγία στη διατύπωσή της δεν ήταν υποχρεωτικά εύληπτη και σαφής στα προβλήματα τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη είναι το θέμα της τεχνολογικής αμεροληψίας ή ουδετερότητας. Επανειλημμένα έχει αναφερθεί αυτό. Δεν πρέπει να προκαθαρίσουμε κομμένες και αραμένες προδιαγραφές που θα ισχύουν. Πρέπει να έχουμε την ελαστικότητα για το δημόσιο τομέα, πώς θα ψηφιοποιεί και πώς θα δραστηριοποιείται. Από την άλλη πλευρά φυσικά να υπάρχει η δυνατότητα εξαιρέσεων Γι' αυτό να υπάρχει αμεροληψία από πλευρά τεχνολογικών εφαρμογών, ώστε να δούμε πώ μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και για το θέμα τη ε, συρρήκνωση του γραφειοκρατικού βάρου και αν θα υπάρχει αρμόδια αρχή, η τροπολογία μου λέει ότι υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες ε, δεν χρειάζεται πάντα να δημιουργούνται νέοι φορείς. Θα πρέπει να δούμε με τους διαθέσιμους πόρους πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίζουν σε αυτόν τον τομέα. Εκεί να γνωρίζουν ποιους πόρους έχουν στη διάθεσή τους και που υπάρχουν οι ανάγκες. Για τα τέλη βλέπω να υπάρχει ανάγκη για τα μουσεία, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και αρχεία ένα μέρος του κόστους τους να μπορούν να το καλύπτουν. Αν στο διαδίκτυο έχουμε τη διάθεση ψηφιοποιημένων αντικειμένων, ε, στοιχείων, που με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα των μουσείων ε, μειώνονται λόγω μειωμένων εισιτηρίων, ε, τότε πρέπει να υπάρχει αντιστάθμιση για αυτές τις απώλειες ε, σε σχέση με τα τακτικά κανονικά τους έσοδα. Στο πεδίο των γενικών δαπανών, ούτως ή άλλως σε σχέση με δήμους και κοινότητες τέτοιου είδους ε, ε, δαπάνες όσον αφορά ε, κτηματολόγια ή μητρώα. Εκείνες οι αρχές πρέπει να αποφασίζουν τι πρέπει να γίνεται και για το manpower, το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται <clears throat> όταν χρειάζεται κανείς τέτοιου είδους στοιχεία και όταν έχουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι άμεσα ελέγξιμα και τεκμηριωμένα. Πρώτα να δούμε ποιο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή του, μετά να δούμε πώς αυτά θα πιστοποιούνται και στην αναγκαία ε, νομοθεσία για την πρόσβαση στα ψηφιακά αυτά ε, στοιχεία. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις ε, για την πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα και σε σχέση με την οδηγία PSA. Σε κάποιες χώρες σε μια οδηγία διατυπώνονται όλα αυτά και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συγχέονται τα μεν με τα δε, αλλά θα είναι ξεχωριστά. Ευχαριστώ. the... Κοιτάξτε, δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Κύριε Σβέτσα, να μην θέλετε να πείτε τίποτα. Πολύ σύντομα όμως. Γιατί θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαρκόφσκι. Μιλήσατε. Μιλήσατε, μιλήσατε. Όταν απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ίσως θα μπορούσε για άλλη μία φορά να τοποθετηθεί γι' αυτό. Διακόπτεται το μικρόφωνο. Διακόπτεται το μικρόφωνο. Τώρα με μικρόφωνο. Για το ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι. Γιατί εγώ υπέθετα ότι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι η Google και άλλοι μπορούν ούτως ή άλλως να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Δεν χρειάζονται αυτοί οι μεγάλοι, η Google και οι άλλοι αυτό το νομοθετικό έργο. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει ποιε είναι οι προθέσεις αυτής της πρότασης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα από δύο από τα σημεία όπου η Κομισιό ε, ζητήθηκε να πει κάτι. Καταρχάς, ε, η, η έρευνα που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους αποκλείεται το πεδίο εφαρμογή ε, του κειμένου και η Κομισιό πριν από την, τις καλοκαιρινές διακοπές υιοθέτησε ένα κείμενο και μία σύσταση για αυτές τις πληροφορίες που καθορίζουν, που κάνουν κάποιες προτάσεις και θα ήθελα να τα διαβάσετε τα κείμενα αυτά. Επίσης, συμφωνώ ότι το Google δεν είναι ο μόνος ε, που ωφελείται από την πρότασή μας, διότι εάν πρέπει να, πληρωθεί, να πληρωθούν τα χρήματα, υπάρχουν αυτά. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το δημόσιο αγαθό θα πρέπει να διανύμεται ε, ε ή μη πληρώνοντας τίποτα ή πληρώνοντας ένα πολύ μικρό ποσό. Αυτό το οποίο βρήκαμε και υπάρχει και μία μελέτη που κάνει η Deloitte, βλέπετε ότι οι δημόσιοι φορείς που έχουν αλλάξει το μοντέλο τιμολόγησης ε, και πήγανε από υψηλή ε, χρέωση σε πολύ χαμηλή, γίνεται, εκεί είχαμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και επαναχρησιμοποίηση και για εμπορικούς και για μη εμπορικούς σκοπούς, για, από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή για άτομα τα οποία... Ε, ενδιαφέρονται. Λοιπόν, η ύπαρξη του δικαιώματος επαναχρησιμοποίησης δεν φύγει τα ε, δεδομένα τα οποία προστατεύονται από συγκεκριμένη νομοθεσία και θα και ίσως δεν θα πρέπει να μιλάτε εδώ πολύ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι υπάρχει παράλληλα και μία πρόταση της Κομισιό που ε, προετοιμάζουμε και εκεί θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, οι κανόνες ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εδώ, αυτό εδώ το κείμενο δεν καλύπτει, αν θέλετε, αυτές τις ανάγκες. Τώρα για τα τέλη υπάρχουν εξαιρέσει και αυτό είναι ένα τομέα τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Η Κομισιόν δέχεται την θέση που αφορά τα πολιτιστικά ιδρύματα, διότι διότι ούτως ή άλλως οι δομές τους και οι απαιτήσεις τους είναι διαφορετικές. Και όντως θα πρέπει ε, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για αυτά τα ιδρύματα. Ραφα, Ραφαέλ, δεν μπορώ να σου δώσω άλλο χρόνο, εκτός αν είναι κάτι πιεστικό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν μίλησα σαν σκιώδης εγώ, αλλά τέλος πάντων και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τη χρέωση. Θα ψηφίσουμε 11 Οκτωβρίου τη γνωμοδότησή σου. Μέχρι τότε ε, θα εξετάσουμε τις συμβαστικές ε, προτάσεις και η κυρία Ρούλη έθιξε το θέμα της προστασίας των δεδομένων αλλά ούτως ή άλλως είπαμε ότι αυτό θα εξεταστεί από άλλη οδηγία για τις συμβιβαστικές τροπολογίες θα δείτε ότι πήρα υπόψη μου τις προτάσεις σας κυρίως όσον αφορά την ψηφιοποίηση και το κόστος και πιστεύω ότι η συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα πρέπει να ε, μας καταστήσει όμοιρους εδώ ε, και ευχαριστώ και την Κομισιό για την ε, διεύκρισή τους. Ευχαριστώ και τους Ιρμηνείς που κάθισαν λίγο παραπάνω. Ήταν πολύ παραγωγικό το πρωινό μας. Στις 3 η ώρα θα τα πούμε και η κυρία Πιτικάινεν θα προεδρεύσει σήμερα το απόγευμα. Θα τα πούμε μετά. Ευχαριστώ.